Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ας ξεκινήσουμε παρακαλώ. Πριν περάσω στο χαιρετισμό των σημερινών μας καλεσμένων, να πούμε πρώτα κάποια τυπικά και διαδικαστικά ζητήματα. Η ψηφοφορία του σχεδίου έκθεσης κυρίας Αγγιλέρα με θέμα τις φαρμακούχες ζωοτροφές, το σημείο δηλαδή 7 της της διάταξης. Αναβάλλεται για την 15η Μαρτίου, γιατί συνεχίζεται ακόμα η συζήτηση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και της ε, εισηγήτριας κυρίας Αγγιλέρα προκειμένου να εκπονηθούν κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Γι' αυτό να βάλετε η ψηφοφορία για τις 15 Μαρτίου. Μέσα στην αλλαγή μόνο προτείνω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Να μεταδίδεται απευθεία από το διαδίκτυο η συνεδρίασή μα και έχουμε ε, διερμηνία σε 20 γλώσσε με εξαίρεση εσθονικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και κελτικά. Αύριο θα έχουμε μόνο σε 16 γλώσσε διερμηνία. θεωρώ ότι μπορούμε να εγκρίνουμε και τα πρακτικά των προηγούμενων μας συνεδριάσεων της 3ης Δεκεμβρίου, η Ιανουαρίου, 18ης και 25 η Ιανουαρίου 2016. Δεν βλέπω αντιρρήσεις, οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά των ε, συνεδριάσεων που προανέφερα. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 4 της ημέρησης διάταξης που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με τον ε, πρώην Επίτροπο, τον κύριο Φραντς Φίσλερ και νυν Πρόεδρο της Διευθύνουσας Επιτροπής του Επιστημονικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διεθνή Έκθεση του Μιλάνου του 2015. Επίσης θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων και με τον David Wilkinson που είναι γενικό εντεταλμένος για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής στη Διεθνή Έκθεση Μιλάνου 2015. Το θέμα της ανταλλαγής απόψεων είναι τα επιτεύγματα της Διεθνούς Έκθεσης Μιλάνου του 2015, της ΕΞΠΟ στο πλαίσιο και των μελλοντικών προκλήσεων της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας γεωργίας. Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω στη συνεδρίασή μας τον πρώην Επίτροπο Γεωργίας και είναι, όπως σας είπα, πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής ε, Διευθύνωσης Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έξπο του Μιλάνου του 2015 με ιδιαίτερη χαρά θα ακούσουμε τα πορίσματα αυτής της Επιστημονικής Επιτροπής στην οποία προεδρεύεται και θα μας παρουσιάσει και κάποιες προτάσεις για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις γνώσεις και τις εμπειρίες που συγκεντρώσαμε από την Expo του Μιλάνου του 2015 για να εξασφαλίσουμε επισητιστική και διατροφική ασφάλεια. Είπαμε ότι έχουμε ε, στη συνεδρίαση και τον κύριο Γουίλκινσον που είναι ο Γενικό Συνδεταλμένο ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ΕΞΠΟ του 2015. Θα μα μιλήσει για τα επιτεύγματα τη ΕΞΠΟ. Ο ε, πρώην Επίτροπο θα μας κάνει μια ενημέρωση για τα πορίσματα της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής μάλλον πρώτα ο κύριος Βίλκινσον για τα επιτέματα της Expo. και μετά ο Επίτροπος Φίτσλερ, πρώην Επίτροπος ε, Φίτσλερ. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψε με τους δύο καλεσμένους μας. Παρακαλώ. Ε, το λόγο έχει πρώτα ο Γενικός Συνδεδελμένος Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή της στην Expo. Ευχαριστώ πολύ. Θα καθίσω στην άκρη για να μπορώ να χειριστώ και τον υπολογιστή, παρακαλώ. So, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to... Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σας σήμερα για να σας δώσω ορισμένα στοιχεία και πληροφορίες για την Διεθνή Έκθεση του Μιλάνου το 2015 από πλευρά και σκοπιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω, το βασικό υλικό θα είναι, εννοείται, η παρουσίαση του κυρίου Φίσλερ ε, σχετικά με τα συμπεράσματα και αποτελέσματα τη Διευθύνουσα ε, Επιτροπή. Όμω, να σα δώσω κάποια κύρια στοιχεία σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μα ε, στο σύνολό τη. Πρώτα απ' όλα, με χαρά μπορώ να πω ότι είχαμε 657.000 επισκέπτες ε, στο περίπτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα στο πλαίσιο, πρέπει να πω, μια ε, εξαιρετικά καλά οργανωμένης ε, εκδήλωση από τι τελικέ Αρχέ. Έκαναν μια τρομερή δουλειά σε ό,τι αφορά ιδίω την ασφάλεια και την προστασία των παρευρισκομένων. Και πρέπει να το αναφέρω αυτό γιατί δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να παίρνουμε για δεδομένο. Όμω πραγματικά ήταν εξαιρετική η διοργάνωση τη έκθεση και ω εκ τούτου με μεγάλη μα χαρά είδαμε ότι ήταν τεράστια και η συμμετοχή των επισκεπτών στο δικό μας περίπτερο. Παράλληλα, είχαμε και πάνω από 250.000 άτομα μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και ιδίως ό,τι φορά τα δικά μας, τις δικές μας σελίδες ε, δικτύων ε, κοινωνικής δικτύωσης ε, ήταν τεράστια συμμετοχή. Πάνω από 50% των συμμετεχόντων ήταν εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την παρουσίαση που είδαν και πάτησαν και το κουμπάκι κατά 95% που είπαν ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι και πάνω από 90% ήταν είτε πολύ ικανοποιημένοι είτε ικανοποιημένοι. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι στο περίπτερό μας είχαμε νέους εθελοντές, ε, φοιτητές του γράμματος Εράσμους από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από 40 χώρες είχαμε φοιτητές. Και πραγματικά η εικόνα που έδωσαν ήταν ε, πολύ θετική και επαγγελματική και για μένα ήταν μία από τις ε, πολύ μεγάλες επιτυχίες σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας. Τώρα, πώς προετοιμάσαμε τη συμμετοχή μας. Θα θυμάστε κάποιοι από εσά ε, στα τέλη του 2013 το Κοινοβούλιο συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει μια κοινή παρουσίαση των δραστηριοτήτων μας. Και από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και εγώ από την Επιτροπή και οι συναδελφοί μου από την Κομισιόν συνεργάστηκαν πολύ στενά με το Κοινοβούλιο, ιδίω ε, το Γραφείο Επικοινωνία στο Μιλάνο και ο Μπρούνο Μελεσάρ που είναι και εδώ και σήμερα. Έκαναν ε, τρομερή δουλειά για την υποστήριξη αυτή τη ε, δραστηριότητα. Συνεργαστήκαμε με 22 γενικέ διευθύνσει πολιτική από την Κομισιόν, εγώ από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο από Επιστημονική Σκοπιά, αλλά είχαμε 22 γενικέ διευθύνσει πολιτική που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί έτσι μπορούμε να δώσουμε ένα πραγματικό ενιαίο ευρωπαϊκό μήνυμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι κατακαιρματισμένα από διάφορε μονάδε και διευθύνσει. Και από το Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Πεφεριών και πολλοί αρμόδιοι φορεί, ιδίω ό,τι αφορά την επιστηστική ασφάλεια και τον αρμόδιο οργανισμό στην Πάρμα. Βεβαίως, ε, πολύ στενή συνεργασία και με του Ιταλούς συναδέλφου που διοργάνωσαν την έκθεση. Αλλά είχαμε και ένα μικρό ρόλο σε... και νομίζω τελικά 19 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαν στην έκθεση. Υπήρξε ένα συντονιστικό έργο και με ένα σύνολο των ε, Γενικών Επιτρόπων από τα κράτη-μέλη. Για να πω οι χώρες που δεν συμμετείχαν είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το περίπτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλέ από τις εκδηλώσεις που ήθελαν να διοργανώσουν, παρότι δεν είχαν δικό τους περίπτερο. Το πιο σημαντικό είναι ότι φτιάξαμε και την ε, Επιστημονική Επιτροπή και θα σα τα πει και ο πρώην επίτροπο. και μαζί με τον Τζαν Κάρλο Καράτη συστήσαμε την ε, Task Force που ε, διεκπεραίων τις καθημερινές μας ε, υποχρεώσεις. Και πραγματικά ήταν πολύ σημαντική δουλειά αυτή για την προετοιμασία και υλοποίηση αυτής της συμμετοχής. Ορισμένα βασικά μηνύματα που συγκρατούμε. Πρώτον, ε, προσπαθήσαμε να έχουμε μια διαφορετική επικοινωνία με το ευρύ κοινό σε σχέση με το παρελθόν. Σε προηγούμενες εκθέσεις, η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν μια πιο γραφειοκρατική ας πούμε, προσέγγιση. Προσπαθήσαμε εμεί να ξεφύγουμε εντελώ από αυτό το πλαίσιο με μια εντελώ διαφορετική προσέγγιση ε, επικοινωνία με το κοινό. Και νομίζω και με μεγάλη ικανοποίηση μπορώ να πω ότι πολύ καλά τα πήγαμε. Είχαμε και ένα καρτούν, μία μικρή ταινία γενομένων σχεδίων, αλλά συμφωνήσαμε και με το βασικό μας μήνυμα. Δηλαδή, συγκεράσαμε παραδοσιακές και καινοτόμες ε, ε, προσεγγίσεις και διαδικασίες. Ε, είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ γεωργίας και επιστήμης, άμα θέλουμε να πετύχουμε τις προκλήσεις μας. Και νομίζω ότι ήταν καλά τα αποτελέσματα. 75% των επισκεπτών τους οποίους ρωτήσαμε ε, μετά, όταν επισκεφθήκαν το περίπτερό μας, είπαν ότι ήθελαν να μάθουν περισσότερα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική για την επιστημική ασφάλεια και 61% των επισκεπτών είπαν ότι η γνώμη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βελτιωθεί. Και πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη ότι βεβαίως ε, οι περισσότεροι από τους επισκέπτες στο περίπτερο ήταν και φιλοευρωπαϊστές. Καλό θα ήταν να έρθουν και κάποιοι πιο ευρωσκεπτικιστέ για να τους εξηγήσουμε ακριβώ τι κάνουμε. Όμω, όσοι ήρθαν είπαν ότι η γνώμη τους φεύγοντα το περίπτερο ήταν ε, πιο θετική. Πρόκειται για μια διοργανική επιτυχία και αυτό είναι κύριο στοιχείο. Ότι παρουσιάσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση από την οπτική γωνία όλων των ε, θεσμικών οργάνων. Ευθύ εξ αρχή ξεκινήσαμε με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, κύριο Μαρτίν Σούλ, μαζί και με την ε, αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Φοντερίκα Μοκερίνη. Ήρθαν, έκαναν τα εγγένεια ε, του περιπτέρου ε, και όλα ξεκίνησαν με πολύ θετικό στίγμα. Τα μισά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ορισμένα αντιπρόσωποι παρευρέθησαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης 85 ευρωβουλευτές συμμετείχαν και επισκέφθηκαν το περίπτερό μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό πλευρά πλευράς διοργανικής επιτυχίας. Πέντε κοινοβουλευτικές επιτροπές, τις βλέπετε εδώ στο, στη διαφάνεια, 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, οι υπουργοί από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και διοργανώσαμε 230 διαφορετικές εκδηλώσεις, φόρα, συναντήσεις πολλών ειδών με συνολική συμμετοχή 30.000 διεθνών εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο για να συζητήσουμε, και να εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα της επιστημιστικής ασφάλειας από όλες τις πτυχές γωνίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, συναντήσεις business to business μεταξύ επιχειρήσεων και η έκθεση είχε πολύ σημαντικό ρόλο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρές στο περίπτερό μας είχαμε περίπου 3.000 διαφορετικές τέτοιε συναντήσει business to business κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου με 1.800 μικρομεσαίε επιχειρήσεις, ομίλους, οργανώσεις τη Ευρωπαϊκή Ένωση με 57 τρίτες χώρες. Κάποιες μεγάλες, κάποιες μικρές. Βλέπετε εδώ και σε έναν ε, κατάλογο του βασικού μα εταίρου και έχουν ήδη συναυθεί 90 συμφωνίες συνεργασίας και πάνω από 700 συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις έχουμε αυτή τη στιγμή. Και ποσοστό ικανοποίηση από τις εκδηλώσεις 85%. Τώρα, πριν δώσω το λόγο στον Φραντ Φίσλερ για να μας ε, μιλήσει για τα πραγματικά επιστημονικά συμπεράσματα από την έκθεση και τι είδους κληροδότημα αφήνει η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Διεθνή Έκθεση. Είναι ένα μικρό βιντεάκι τώρα που φτιάξαμε στο τέλος για να έχετε μια γενικότερη εικόνα. Ε, θα καλέσω τον τεχνικό να έρθει να με βοηθήσει. Okay,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 sforzo di comprensione e innovazione a livello globale. Okay, so thank you very much, ladies and gentlemen. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα τον λόγο στο Φραντς Φίσλερ. Κύριε Πρόεδρε, Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε δυνατότητα να σας παρουσιάσω τη δουλειά της ε, Διευθύνης Επιτροπή. Επιτροπής. Ε, δουλέψαμε δυόμιση χρόνια και έχουμε ε, εκδώσει και μια, ένα ενημερωτικό φυλάδιο που μπορείτε να το βρείτε βγαίνοντα από την αίθουσα. Μπορείτε λοιπόν, όπως σας είπα, να πάρετε ένα αντίτυπο Η πρωτοβουλία να συσταθεί αυτή η Διευθύνουσα Επιτροπή, η πρωτοβουλία αυτή ανελήφθη από κοινού, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την τότε Ιταλική Προεδρία. Η ιδέα δεν ήταν τίποτα άλλο από το να πούμε και να προβάλλουμε ότι η Ευρώπη οφείλει να είναι ένας από τους βασικούς παίκτες ε, στο ερώτημα τι ακριβώς πρέπει να γίνει έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη να έχουν ε, επάρκεια τροφίμων. Η παγκόσμια ε, συντηστική επάρκεια, αυτή ακριβώς ήταν το θέμα και ξεκινήσαμε μισό λεπτό. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μια στρατηγική έρευνα και εντοπίσαμε πρώτα απ' όλα μια ε, στρατηγική προσέγγιση και αυτή η στρατηγική προσέγγιση είναι ένα είδος ε, εικονικού ελικοειδούς που πρώτα απ' όλα εντοπίζει στους ε, τομείς όπου πρέπει να γίνει έρευνα, μετά γίνεται η έρευνα και κατόπιν τα αποτελέσματα της έρευνας ε, είναι εκείνα που αποφέρουν τη γνώση. Και μετά είναι απαραίτητο να υπάρξει και άλλη μια αλλαγή έτσι ώστε τα απορίσματα της έρευνας να μεταφραστούν σε νέες τεχνικές, νέες τεχνολογίες και με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να επιτύχει ε, κάποια, να ασκήσει επιρροή σε κοινωνικό επίπεδο και μετά να υπάρξει πρόοδος. Και ε, αυτή η διαδικασία να έννοει. Συνειδητοποίησαμε λοιπόν επτά τομείς προτεραιότητας για την έρευνα. Δεν νομίζω βέβαια ότι χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά αυτούς τους ε, τομείς, αλλά θέλω να σας πω ότι καλύψαμε όλα τα θέματα που κατά την άποψή μας είναι σημαντικά. Αν θέλουμε βέβαια να υπάρχει επάρκεια τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευτής εξ αρχής ταχθήκαμε υπέρ μιας ε, αηφόρου αποκαλούμενης διαδικασίας. Δηλαδή το δικό μας το σχέδιο ταιριάζει θαυμάσια και με τις νέες μορφές STG όπου μπορεί κανείς να συνδυάσει και την οικονομία και την οικολογία μεταξύ άλλων. Κατόπιν, ναι, Κατόπιν κλήθησαν όλοι να συμμετάσχουν σε αυτή την πρόκληση και καταλήξαμε σε τέσσερις συστάσεις. Βλέπετε λοιπόν τι ακριβώς συνιστούμε. Συνιστούμε πρώτα απ' όλα το εξής. Το καθήκον μας δεν είναι να ε, στηρίξουμε μια νέα πολιτική, αλλά μια ερευνητική προσέγγιση. Επίσης, η στόχη μας, ή το καθήκον μας, ε, είναι όλα αυτά τα συστήματα από τον αναλυτικό τομέα να τα εντάξουμε μέσα σε ένα σύστημα. Σημασία έχει επίσης να αλλάξουμε ε, με τον ίδιο τρόπο και την προσέγγισή μας. Η έρευνα ε, κατατμείται, κατακαιρματίζεται σε διάφορους υποτομείς. Κάθε ένας ε, από αυτούς τους υποτομείς είναι σαν μία αποθήκη, σαν ένα σιλό και αν όμως συνεχίσουμε τον τρόπο αυτό δεν θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε τα διάφορα στοιχεία και να επιτύχουμε το στόχο μας που είναι ψηφιστική ασφάλεια. Άρα δηλαδή το πρώτο που συστήνουμε είναι να εξετάζουμε συστημικά το όλο θέμα, δηλαδή να αντιμετωπίζεται το μέσον τροφίμων ως ένα πολύ περίπλοκο σύστημα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος για να ξεφύγουμε από αυτήν την ε, προσέγγιση. Η σύσταση υπαριθμών 2 είναι στράτευση. Άρα δηλαδή όλα τα τμήματα της κοινωνίας πρέπει να ενταχθούν μέσα σε αυτή την πρόκληση ε, που αφορά στα τρόφιμα και τότε οι ερευνητές, οι πολιτικοί, οι οικονομολόγοι, οι ΜΚΟ και πολλοί άλλοι, μόνο αν όλοι αυτοί συνδυαστούν, μόνο τότε ε, θα προκύψει μια καλύτερη ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να δοθεί όθηση και στην καινοτομία. Τέταρτη σύσταση, τέσσερις υποβάλαμε. Η τέταρτη σύσταση αφορά σε ένα διεθνές πάνελ για την συντηστική και διατροφική ασφάλεια. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Βλέπετε λοιπόν και πάλι αυτούς τους επτά τομείς ε, ε της... Ε, πρωτοβάθμιας έρευνας ε, που είναι απαραίτητη και όπως σας είπα η πρώτη σύσταση είναι όλα αυτά που προνέφερα να συνδυαστούν. Δηλαδή αυτή η υποτομή και η έρευνα σε αυτούς όλα αυτά να συνδυαστούν. Αυτό κατ' ουσίαν σημαίνει συστημική προσέγγιση και επίσης και διατομεακή έρευνα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να μετατρέψουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας σε πρακτική εφαρμογή, να τα χρησιμοποιήσουμε στην πράξη, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ασκήσουμε επιρροή. Όσο τα αποτελέσματα, τα πορίσματα της έρευνας δημοσιεύονται μόνο σε επιστημονικές, πανεπιστημιακές μελέτες και δεν εφαρμόζονται στην πράξη, ε, παραμένουν ε, χωρίς αποτέλεσμα. Ό,τι κάνουμε δεν έχει άμεση απήχηση. Η τρίτη μας σύσταση είναι να επιτύχουμε ένα καλύτερο περιβάλλον καινοτομία. Ας δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Αν λοιπόν επιθυμεί κανείς να επιφέρει καινοτομίε, είναι σαφές ότι χρειάζεται νέες ιδέες, αλλά δηλαδή χρειάζεται και νέα έρευνα. Και κατόπιν πρέπει κανείς να προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα και από τα πορίσματα της έρευνας ε, να καταλήξει νέες έρευνες. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται όμως κανείς και τον επιχειρηματικό κόσμο, τους επενδυτές οι οποίοι από αυτά τα πορίσματα καταλήγουν σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Και για να γίνουν αυτά χρειάζεται κανείς επενδυτικά κεφάλαια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ε, καινοτομία και σχετική περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία περιλαμβάνει και την επικοινωνία. Οι πολίτες μας ε, πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τι ακριβώς ε, εννοούμε όταν μιλάμε για καινοτομία και γιατί όλα αυτά τα οποία προγραμματίζουμε είναι καλά για τις κοινωνίες μας γενικά, για τις κοινωνίες όλου του κόσμου και όχι μόνο στη δική μας την πατρίδα. Βλέπετε λοιπόν εδώ στη διαφάνεια και τους κύκλους οι οποίοι οδηγούν, όλοι αυτοί οδηγούν στην αηφορία. Αηφορία σημαίνει αυτό το τρίγωνο που αποτελείται από οικονομία, οικολογία και κοινωνική ευθύνη. Τώρα πάμε στην τέταρτη σύσταση. Γνωρίζετε όλοι σας ότι υπάρχει ένα διεθνές ε, πάνελ, ένα βήμα συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή. Εμείς λοιπόν σκεφτήκαμε ότι δεν θα ήταν άσχημο να αναζητήσουμε τρόπους για το πώς μπορούμε κάτι παρεμφερές να το εισάγουμε και στον τομέα των τροφίμων. Τα τρόφιμα είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί στον πλανήτη μας εξακολουθούν να υπάρχουν 800, 800 εκατομμύρια άνθρωποι που υποφέρουν από πείνα ή κακή διατροφή. Αξίζει λοιπόν τον κόσμο να σκεφτεί κανείς ε, ένα τέτοιο θεσμό, γιατί πρώτα απ' όλα αυτός θα μας επέτρεπε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία ανάμεσά μας και δεύτερον θα μας ε, έδινε τη δυνατότητα να προβαίνουμε σε ε, αξιολογήσεις, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να κάνουμε έλεγχο, να διαπιστώνουμε κατά πόσον σημειώνουμε πρόοδο και όχι. Αν δει λοιπόν κανείς λιγάκι τη δομή αυτού του πάνελ, τουλάχιστον στον τομέα της ε, κλιματικής αλλαγής, πρόκειται για ένα συγκερασμό ανάμεσα σε πολιτικούς και επιστήμονες. Παράλληλα όμως είναι και ένας ε, συμβιβασμός ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Ε, την καθοδήγηση την, έχει ο, την έχουν οι πολιτικοί και όχι τόσο οι ερευνητές. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, προτείναμε τρεις δυνατότητες. είτε να ακολουθήσουμε ε, το ίδιο μοντέλο όπως την κλιματική αλλαγή ή να το αλλάξουμε λιγάκι, δηλαδή να ε, δώσουμε περισσότερη σημασία, να δώσουμε το πρώτο χέρι στους ε, επιστήμονες και όχι στους πολιτικούς. Ή αν θέλετε μπορούμε να συνεχίσουμε με το σύστημα ως έχει και αυτό βέβαια σημαίνει ότι ο έλεγχος που προβλέπεται από τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο των στόχων της ε, αηφόρου ανάπτυξης ε, δεν θα επιτευχθεί. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω το εξής. Η πολυτομεακή έρευνα είναι εκείνη που κάνει τη διαφορά, που σημαίνει και συνεργασία ανάμεσα στους ερευνητές. Υπερτομεακή, η διατομεακή συνεργασία σημαίνει τα πορίσματα των επιστημόνων να υιοθετηθούν από το βιομηχανικό κόσμο, από τους πολιτικούς και από τους πολίτες. <coughs> Πρέπει λοιπόν και εμείς να συμβάλλουμε και αυτή είναι μία πρόσκληση που απευθύνω σε όλους σας. Σας καλώ να μην ε, παραγνωρίζετε τη σημασία της ε, συντηστικής ε, ασφάλειας. Γιατί ας ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο γύρω μας, ας δούμε τι συμβαίνει στη Συρία και στους καταβλισμούς προσφύγων ή στην Ανατολική Αφρική. Η επισητιστική ασφάλεια είναι όλο και περισσότερο ένα κρίσιμο θέμα. Αν λοιπόν στο μέλλον δεν κατορθώσουμε να έχουμε τρόφιμα για όλους, δεν θα επικρατήσει και ποτέ ειρήνη στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. για τις παρουσιάσεις, κύριε Βίλκινσον, κύριε Θίσλερ. Διαμορφώσατε ένα πλαίσιο ε, για τις περαιτέρω ενέργειες που θα μπορούσαμε να αναλάβουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διδάγματα που αντιλήσατε και τα πορίσματα από τη Διεθνή Έκθεση του Μιλάνου για το 2015. Ξέρετε ότι ο κ. Δεκάστρο ήταν επικεφαλής ε, της ε, αντιπροσωπείας μας ε, για την ΕΞΠΟ και επίσης συμμετείχε και στην διοργάνωση. Παρακαλώ κύριε Δεκάστρο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Βεβαίως θέλω να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα ευχαριστώντας όχι μόνο τους δύο μιλητές μας, τον κύριο Φίσλα και τον κύριο Βουίλκινσον, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των ε, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολύ καλή δουλειά τους. Συνέστησαν μια διευθύνουσα επιτροπή που δούλεψε πάρα πολύ τους ε, τελευταίους πίνες. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω πρώτα απ' όλα το εξής. Να μην χαθεί αυτή η πάρα πολύ καλή δουλειά που έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια των έξι μηνών της ΕΞΠΟ. Οι αριθμοί που μας παρουσίασε ο κύριος Γουίλκινσον ε, μιλάνε από μόνοι τους, ε, ε, μεγάλη επιτυχία της ΕΞΠΟ και πάνω από 21 εκατομμύρια επισκέπτες. Ευχαριστώ βεβαίως και την δουλειά που έκαναν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και εγώ θα ήθελα να καλέσω όλους τους συναδέλφους να διαβάσουν αυτό το ενημερωτικό φυλάδιο που μας έδωσε ο κύριος Φίσλερ. Εκεί λοιπόν περιλαμβάνονται και τα ε, συμπεράσματα όλης αυτής της δουλειάς γιατί πραγματικά εγώ είμαι εντυπωσιασμένο από όλη αυτή τη δουλειά που έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δύο πράγματα θέλω να πω. Το είπε και ο επίτροπο κ. Φίσλερ. Καταρχήν ε, το θέμα ε, τη επισητιστική ασφάλεια, που είναι ένα θέμα παγκόσμιο. Εάν λοιπόν ε, θέλουμε να προβάλλουμε λιγάκι το τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόρθωσε να ευαισθητοποιήσει για την πρόκληση ευαισθητοποίηση λοιπόν για το ότι είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε τη σωστή κατεύθυνση, να υιοθετήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της ε, διεπιστημονικής και διατομεακής έρευνας και συνεργασίας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα συμπεράσματα ε, προέκυψαν από τη δουλειά της Επιτροπής ε, Juncker και Θέλω επίσης ε, να σας πω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον ε, Μπανκιμούν. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ε, κύριος Φίσλερ, έστειλε μια σχετική επιστολή και εκεί αναφέρεται αυτή η δουλειά από πλευρά Ηνωμένων Εθνών, οι εντυπώσεις που άφησαν συγκεκριμένες προτάσεις κάτι που ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος κ. Γιούγκερ θα το αφήσει να χαθεί, αλλά θα το χρησιμοποιήσει στις επόμενες ε, μεγάλες ε, συναντήσεις του. Ε, θα γίνει ας πούμε στο Καζακστάν σύντομα μία συνάντηση στον διάμεσο χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη έξπο που θα γίνει το 2020 στο Ντουμπάι. Όσον αφορά την αηφορία και κλείνω με αυτό, ε, θέλω να απογραμμίσω αυτά που μας είπε ήδη ο Επίτροπος κ. Φίσλερ, δηλαδή η αηφορία, η αηφόρος ανάπτυξη και η επισητιστική ασφάλεια. Αυτά είναι δύο θέματα που πρέπει να τα επαναξετάσουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προσφέρουμε τρόφιμα σε όλους τους κατοίκους που αλλάζουν διατροφικές συνήθειες. Οι πολίτες οι άνθρωποι επιθυμούν όλο και περισσότερα τρόφιμα, άρα δηλαδή πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερη σημασία και στην έρευνα και στην καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους δύο τομείς κάνει πάρα πολλά, αλλά ίσως ε, δεν κάνει αυτά που είναι απαραίτητα. Για άλλη μια φορά λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την ομάδα που εργάστηκε για την έκθεση και να σας συγχαρώ για την εντυπωσιακή προσφορά σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς κύριε Δεκάστρο και σας ευχαριστούμε για την μεγάλη συμβολή σας στις εργασίες της συναφής με την Expo και το έργο σας και για το μέλλον και τις πρωτοβουλίες που θα λάβετε στο μέλλον. Ο κύριος σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής και τον κύριο Φραντς Φίσλερ. Η έκθεση για την Expo στο Μιλάνο, από αυτού θέλω να πω ότι εγώ δεν ήμουν ένας από τα 21 εκατομμύρια επισκέπτες, όμως ε, παρακολούθησα εξ αποστάσεως. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μία απόφαση για την ΕΞΠΟ και διάβασα κάποια σημεία αυτή τη έκθεση. Αναφέρεται λοιπόν το εξή. Για να καταστεί δυνατόν στι γεωργικέ επιχειρήσει να υπάρξει αεφόρο ανάπτυξη, γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί πέφτουν οι τιμές των προϊόντων μας ε, το δικαίωμα σε τρόφιμα είναι ένα θεμελιώδη δικαίωμα των ανθρώπων και γι' αυτό καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει τρόφιμα στον πλανήτη. Ο κύριος Φίσλε το είπε ότι έχουμε 800 εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη μας που δεν έχουν να φάνε. Ε, δηλαδή, ναι με μειώθηκε αναλογικά το ποσοστό γιατί αυξήθηκε το σύνολο του πληθυσμού στον πλανήτη, αλλά παρόλα αυτά, αυτά τα 800 εκατομμύρια που δεν έχουν ε, επαρκή τρόφιμα, αυτό δεν μπορεί να υφίσταται, γιατί ο πλανήτης μπορεί να θρέψει όλους τους ανθρώπους. Τίθεται μόνο το θέμα της ε, κατανομής και της παραγωγής. Εγώ από τα 14 μου χρόνια είμαι γεωργός και αυτό που με συγκλονίζει είναι ότι από τα 800 εκατομμύρια ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε πάνω από 500 εκατομμύρια είναι μικροί γεωργοί. Άρα δηλαδή δεν επιτρέπεται οι γεωργοί οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ένα ή ενάμιση εκτάριο, οι άνθρωποι αυτοί ε, να μην έχουν τις πρώτες ύλες, να μην έχουν τους σπόρους, να μην έχουν την τεχνολογία, να μην έχουν το νερό και γι' αυτό να πεινάνε. Εγώ έχω πάει στη Βραζιλία ε, που είναι γεωργική χώρα και αν δει κανεί ε, το πόσο πεινάνε οι άνθρωποι εκεί, πραγματικά ε, συγκλονίζεται. Ελπίζω λοιπόν μετά την έξπο του Μιλάνο να υπάρξει κάποια συνέχεια. Μιλάμε για υφόρο ανάπτυξη στην Γεωργία. Ελπίζω να συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση η έξπο και ο κύριος Φίσλερ πολύ σωστά είπε ότι η έρευνα πρέπει να οργανωθεί καλύτερα. Γνωρίζω πολύ καλά η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχει ένα ομοσπονδιακό σύστημα διακυβέρνησης με 16 κρατήδια και στη Γερμανία τη δεκαετία του 70 ή και το αργότερο ε, μετά την επανένωση ε, δεν ζητούσαν ε, και δεν ερευνούσαν όλα τα κρατήδια το ίδιο πράγμα. Άλλα ερευνούσε το ένα, άλλα ερευνούσε το άλλο. Φανταστείτε λοιπόν σε μία και μόνο χώρα εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερο συντονισμό των ερευνητικών προσπαθειών, καλύτερη χρήση των κονδυλίων, γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα το πρόβλημα της επιστημιστικής ασφάλειας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε η έξπο στο Μιλάνο και όπως είπε και ο συνάδελφος κύριο Ντεκάστρο, που ασχολήθηκε πάρα πολύ. Η έκθεση αυτή ε, άφησε τη σφραγίδα της και αυτή η σφραγίδα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε στο μέλλον να υπάρχει καλύτερο συντονισμός. Το ε, πρόβλημα το προσφυγικό έχει άμεση σχέση και με την επισητιστική ανεπάρκεια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε όλοι από κοινού τι πρέπει να κάνουμε για να ελέγξουμε το πρόβλημα στη Βαβαρία έλαβε χώρα η συνάντηση των G7 και εκεί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είπαν ότι μέχρι το 2030 ε, θα πρέπει να ε, μειωθεί στο ίμιση ο αριθμός των ανθρώπων που θα πεινάνε. Εγώ λέω μέχρι το 2030 να μην πεινάει πλέον κανείς. Ήδη σήμερα μπορούμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα με βάση το οποίο ε, θα έχουμε στόχο, όπως σας είπα, να έχουμε ε, ως ανθρώπους με πρόβλημα διατροφής 400 εκατομμύρια. Εγώ δεν συμφωνώ, κανείς να μην πεινάει, κανείς να μην έχει ανάγκη επισητιστικής βοήθειας και οι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν εκεί που μεγάλωσαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο και ευχαριστώ επίσης ε, και τους εμπειρογνώμονες ε, για το ότι μας δίνουν δυνατότητα να δούμε λιγάκι αναδρομικά την ΕΞΠΟ. Και εσένα Παόλο Ντεκάστρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ασχολήθηκες πολύ με την ΕΞΠΟ, το σεβασμό μας, υποκλεινόμαστε ε, αυτά ε, είχαν αποσθετικά, τώρα δεν ακολουθήσουν και τόσο θετικά. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ΕΞΠΟ και δικαίως εμφανίστηκε στον κόσμο ως μια έκθεση που δεν ήταν ε, απόλυτα συνδεδεμένη με θετικές εξελίξεις. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα έχουμε κατά νου, πρέπει να τα εξετάσουμε. Εγώ ξέρω το τι ελέγχθη στη Γερμανία αλλά και σε άλλες εφημερίδες διάβασα κριτική σε σχέση με την έξω. Μα πώς είναι δυνατόν το Βατικανό, το θέμα της πείνας, να είναι το Βατικανό εκείνο που να φέρνει το θέμα αυτό επιτάπητος. Πώς είναι δυνατόν οι φτωχότερες χώρες του κόσμου ε, να μην μπορούν να συμμετέχουν στην έξπο. Πώς είναι δυνατόν όμιλοι επιχειρήσεων που ρυθμίζουν όλα αυτά ε, να μην εκφράζουν κανένα σχόλιο. Το θέμα της ε, διαφυγής από εμπόλεμες περιοχές ε, αυτό δεν έχει σχέση με τους πρόσφυγες στη Γερμανία στην Ευρώπη. Αυτό έχει γενικά με τη διαφυγή, ένα είδος διαφυγής που ζούμε εδώ και δεκαετίες. Φεύγουν άνθρωποι μέσα στις πατρίδες τους, δεν μπορούν πια να μείνουν στα χωράφια τους. Βλέπουμε από την τηλεόραση ε, διάφορες καταστάσεις, αλλά τελικά δεν γίνεται τίποτα. Εσείς λοιπόν είστε υπεύθυνοι και γι' αυτό οφείλετε να επιληφθείτε και αυτών των αρνητικών εξελίξεων σε σχέση με την Expo. Αυτό που μας είπατε είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη αλήθεια, η άλλη μισή είναι ότι η Coca-Cola, η Nestlé και άλλοι είχαν μια πλατφόρμα για να διαφημιστούν. Και ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει η Nestlé με την κατασκευή πηγαδιών. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεχίσουν να ασχολούνται με τη Γεωργία γιατί τους παίρνει το νερό, είναι στυλά για τα πηγάδια της. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν ε, και οι πολυεθνικές αυτέ αυτές τις αλλά είμαστε υποχρεωμένοι όταν μιλάμε να μιλάμε ειλικρινά και να μην τα παρουσιάζουμε όλα τέλεια. Κάτι άλλο, η Ευρώπη δεν έχει το καθήκον και δεν είναι δουλειά της να τρέψει όλο τον κόσμο. Η Ευρώπη όμως οφείλει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να τραφεί μόνος του. Να ε, πάρουμε τα χέρια μας πίσω από αυτούς που, στα, που τους τα αρπάζουμε. Εντάξει, στην Expo έγιναν καλές συναντήσεις, ε, δείξατε το θέμα της έρευνας, ε, δεν το αμφισβητώ, αλλά η Expo έχασε μία μοναδική ευκαιρία να δώσει κίνητρα για να σκεφτούμε συζητούμε και να ξανασυζητηθεί το θέμα της διατροφής σε παγκόσμια κλίμακα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Άγνιο. Μέχρι πριν από μία ώρα κάποιος με ρωτούσε ε, γιατί έγινε η έξοδο του Μιλάνου. Θα το απαντούσα όταν ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο της ε, ε, Ιταλική κυβέρνησης για να προβάλλει την Ιταλία στην Ευρώπη και στον κόσμο με όλα τα καλά προϊόντα που παράγει η χώρα αυτή και να προσελκύσει ερευνητές από όλες τις χώρες του κόσμου γιατί στη Βόρεια Ιταλία έχουμε αναγνωρίσει ότι είναι πραγματικά ένα κόμβος καινοτομίας. Μετά όμως, μία ώρα μετά και βλέποντας ε, και το βιντεάκι αυτό, βλέπω ότι ήταν μια τεράστια προπαγανιστική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου τα χαλάσατε κάπως γιατί ε, καπηλευτήκατε τις προσπάθειες της τελικής κυβέρνησης και τελικά ε, έτυχε που έγινε η έξω στο Μιλάνο ή στην Ιταλία. Δεν έχει σχέση φαίνεται το αντικείμενο με την Ιταλία. Ένα από τα θέματα της έκθεσης ήταν η πιστιστική ασφάλεια και αναφέρθηκαν 7 σημεία για το πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε το στόχο της επιστηστικής ασφάλειας. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ούτε σε ένα από τα σημεία αυτά δεν αναφέρθηκε η μείωση της εξάρτησης μας από τις εισαγωγέ των τροφίμων. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που όλοι το ξέρουμε και φαίνεται να το αγνοούμε. Γιατί ε, από την Νότια Αμερική εισαγάγουμε χιλιάδες τόνους ε, γενετικώς τροποποιημένης σόγιας γιατί οι Ευρωπαίοι Γεωργοί δεν επιτρέπεται να καλλιεργούν γενετικώς τροποποιημένη σόγια. Και πολλέ ομάδε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να ξυπνήσουν, γιατί τα πράγματα προχωρούν. Θα πρέπει να θετήσουμε νέε τεχνολογίε. Αν δεν το κάνουμε, θα γίνουμε ένα γεωργικό μουσείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πράγματα είναι απλούστατα. Επίση, αναφέρθηκε η συστημική σκέψη, το system thinking. Ποια είναι αυτή η συστημική ε, σκέψη, το σύστημα σκέψης γιατί αν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες αναπτύσσουν μια τεχνολογία ή κάτι, τότε όλα αυτά είναι, φαίνεται να λέτε ότι είναι ε, περιτά αν ε, ε, αποφέρουν μόνο καρπούς για την πολυεθνική ε, εταιρεία. Είμαστε τόσο μυσαλόδοξοι απέναντι στις πολυεθνικές εταιρείες που απαξιώνουμε οτιδήποτε προσπάθεια και αν κάνουν. Κάποιο που έχει επιστημονικό ενδιαφέρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ικανότητε και δεξιότητε και παράγει κάτι χρήσιμο, είναι κρίμα να απαξιώνεται από τους ε, πολέμιους του μόνο και μόνο επειδή είναι κατά των πολυεθνικών. Γιατί τέτοιοι ερευνητέ απλώς ε, θα ε, μεταβούν κάπου αλλού και θα βουλιάξουμε ακόμη πιο πολύ σε αυτή τη μοίρα μας να γίνουμε ένα γεωργικό μουσείο. Και τώρα, για το περιβάλλον. Βέβαια, αν αλλάζει το κλίμα θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους γεωργούς ε, να προσαρμοστούν. Αλλά φαίνεται ότι τις μέρες μας έχει διαφορετική έννοια αυτό, αυτή η έννοια. Φαίνεται ότι ε, συμβάλλουν και οι γεωργοί στην αλλαγή. Ποια από τις δύο εναλλακτικές θεωρείτε ότι είναι σωστή. Σας ευχαριστώ κύριε Άγνιου. Ο κύριος Πέτερλε. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο. Eh, eh. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι μέλος και της Επιτροπής Περιβάλλοντος και επίσης συμπρόεδρος και στην ομάδα εργασίας για την υγεία και μελισσοκόμος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φίσλερ και τον κύριο Γουίλκινσον για τις παρουσιάσεις τους και να τους συγχαρώ για τις δραστηριότητες και τις ενέργειές του στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης του Μιλάνου. Εγώ είμαι από τους ικανοποιημένους ε, της γεωρικής διάστασης που είχε η έξπο του Μιλάνου. Βέβαια, αναφέρθηκαν κάποιες κριτικές από συναδέλφους και μπορεί μερικέ να ευσταθούν, αλλά νομίζω ότι το μήνυμα ήταν θετικό γιατί η συνεργασία μας ήταν αγαστή και επίσης συνάντησα και πολλούς νέους που δεν ήταν πολέμοι της Ευρώπης, δεν ήθελαν λιγότερη Ευρώπη, αντίθετα ήθελαν περισσότερη οικολογία και περισσότερες περιβαλλοντικές ανησυχίες. Νομίζω ότι σήμερα βρήκαμε μια σωστή προσέγγιση και διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε πρόοδο αν δεν έχουμε μια συστημική ενοιολογική προσέγγιση και δεν μπορούμε να επιτύχουμε την βιωσιμότητα αν δεν αναλάβουμε κι εμείς μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί από τους παγκόσμιους εταίρους. Επίσης δεν θα πρέπει να ερμηνεύουμε την πρόοδο μόνο ποσοτικά και το θέμα της επιστηστικής ασφάλειας. Το θέμα δεν είναι πολλά, μεγάλη ποσότητα τροφίμων, αλλά υγιεινά τρόφιμα. Αυτό είναι επιστηστική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Χόιμπους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε η Μαρία. Και εγώ λοιπόν ε, είδα λιγάκι την Expo, πήγα επί τόπου και πρέπει να σας πω ε, η προσέγγιση αυτής της έκθεσης ήταν ε, πολύ τεχνική και πολύ προσανατολισμένη σε ανάπτυξη. Πράσινη ανάπτυξη, στην Ασία. Βεβαίως και τότε προέκυψε ανάπτυξη, αλλά για να δούμε εντωμεταξύ τι ζημιά προέκυψε σε αυτές τις περιοχές. Για να δούμε τι έγινε με τα εδάφη μας, με την ε, υδροδότηση. Για να δούμε λιγάκι πώς άλλαξαν οι κοινωνικές σχέσεις μέσα στην ίδια τη Γεωργία. Και αν δούμε το που πεινάνε περισσότεροι άνθρωποι, είναι ακριβώς σε αυτή την περιοχή. Ε, θέλω λοιπόν να σας πω ότι εμένα δεν μου αρέσει ε, αυτή η προσέγγιση. Κύριε Φίσλα, στο τέλος της ε, παρέμβασής σας ε, είπατε ότι πρέπει να υπάρχει διατομεακή συνεργασία. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας, αλλά εσείς αυτή τη συνεργασία την περιορίσατε μόνο στην επιστήμη. Εγώ πιστεύω ότι αν θέλει κανείς να συνεργάζεται διατομεακά, ε, δεν πρέπει να αφήνει εκτός ε, τους γεωργούς. Πρέπει κανείς να συμπεριλαμβάνει και τη δική τους τη γνώση, να ενημερωθεί κανείς για το ποιες είναι οι ανάγκες τους. Δεν μπορούμε να συστήσουμε επιστημονικά κάτι το οποίο στην κοινωνία δεν υφίσταται. Οφείλουμε να λάβουμε περισσότερο υπόψη μας ε, τις ε, δικές τους τις ανάγκες για να καταλήξουμε σε ανθεκτική παραγωγή. Αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε ε, χωρίς τους γεωργούς απλά και μόνο με επιστημονική προσέγγιση. Για να δούμε λιγάκι τους σπόρους. Υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία πατάτας από τη Γερμανία προς την Κένια, δηλαδή γερμανικές αλλά και ολλανδικές πατάτες αυτές ε, στέλνονται στην Κένια και καλλιεργούνται. Ε, αυτές είναι ε, καλές ποικιλίε για τηγανιτές πατάτες και τσίπς. Όμως δεν είναι τόσο, δεν ενδείκνυνται όπως οι τοπικές ποικιλίε. Αυτό ήταν ένα απλό παράδειγμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι με τέτοιου είδου προσεγγίσεις μπορούμε να προχωρήσουμε. Ε, πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου όλα αυτά που διαδραματίζονται επιτόπου σε μία χώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Τσούλο. E ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τους για γιατί παρουσίασε της δουλειάς τους. Και θέλω να πω το εξή. Ε, συμφωνώ με αυτό που λέτε για τις ε, πρακτικέ ενέργειε. Η πρόκληση της ΕΞΠΟ ήταν να προβληθεί το δικαίωμα στη διατροφή, στα τρόφιμα, ε, όχι μόνο και διατροφή αλλά και με υγιεινό τρόπο. Κάτω λοιπόν από αυτό το πρίσμα είμαι πεπισμένος ότι επιτέθηκε ο στόχος με την έννοια ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή επιτεύχθηκαν αποτελέσματα. Για μας το σημαντικότερο από όλα είναι ότι διατηρήθηκε η διατροφική κυριαρχία. Και επίσης δώσαμε τη δυνατότητα να εκπροσωπηθούν κάποιοι οι οποίοι όμως είναι αρπακτικά για τους αδύναμους. Όσον αφορά τους στόχους που θα έπρεπε να επιτύχει αυτή η πρωτοβουλία, θέλω να ρωτήσω κατά πόσο πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει έναν καθοδηγητικό ρόλο για να διασφαλιστεί το δικαίωμα στη διατροφή. Και αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να το κάνει με τη μορφή του συντονιστή σε διεθνές επίπεδο. Δεν πρέπει η Επιτροπή να περιορίζεται σε ευρωπαϊκά σύνορα. Και αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα, γιατί όσο πιο πολύ χρόνο χάνουμε, τόσο χειρότερα. Το δικαίωμα στη διατροφή είναι κάτι το οποίο αφορά το περιβάλλον, ε, την υγεία. Δεν μπορούμε πια να χάνουμε άλλο χρόνο αν πραγματικά θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο με σοβαρότητα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Φλάναγκαν, ευχαριστώ πολύ για την εγώτα που μου δίνετε να πάρω το λόγο. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε και το βιντεάκι πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι ο σκοπός ε, των όσων μας είπατε ήταν ότι θέλετε κι εμείς ε, να διαβιβάσουμε αυτό το μήνυμα περαιτέρω και να αναλάβουμε και δράση. Παρατήρησα λοιπόν στο βίντεο και δύσκολα μπορεί κανείς να διαφωνήσει με τον βουλευτή Άγνιου ότι ουσιαστικά ήταν ένα προπαγανδιστικό βίντεο όπου μας είπαν όλα αυτά τα ωραία που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ήταν μια φανταστική επιτυχία. Εγώ διερωτώ με. Και μπορείτε να μας πείτε και να σχολιάσετε κάτι ότι και πάλι και σήμερα πολύ λίγοι ευρωβουλευτές ήρθαν εδώ. Ως πολιτικός βέβαια πρέπει κανείς ε, να πάρει αποφάσει για το πού θα παρευρεθεί κάθε μέρα. Αυτό ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα ε, αυτό που μας περιγράφεται σήμερα. Παρ' όλα αυτά οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν και επέλεξαν να πάνε κάπου αλλού. Επομένως, αν αυτοί που έχουν εκλεγεί για να τα, κάνουν, να τα ακούσουν όλα αυτά ε, και δεν έρχονται καν σε αυτή τη συνάντηση, τι ελπίδες έχουμε τελικά για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Δείχνει κάτι για τη σημασία που αποδίδουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σφερού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο στόχος ε, της έκθεσης Μιλάνο 2015 ήταν ε, πραγματικά ε, πολύ θετικός, διασφάλιση της επιστηστικής και διατροφικής ασφάλειας. Δεν έχω τίποτα να πω. Και εγώ μάλιστα πήγα στο Μιλάνο και είδα με τα μάτια μου ότι οι Ιταλοί φίλοι μα πολύ καλά διοργάνωσαν ε, την έκθεση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ζητήματα επί για το Ταμείο ε, παραγωγικότητα ε, και καινοτομία, όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε και η Γαλλία έχουν την καλύτερη δυνατή θέση για αυτό το ζήτημα. Η Γαλλία και οι ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν υπόψη και τις προσπάθειες των πολιτών και τους προβληματισμούς τους με την αρχή της προφύλαξης, ιδίως ό,τι αφορά τα γενετικώς τροποποιημένα, αλλά και τη διατήρηση της υψηλή ποιότητα παραγωγής. Και αυτό και η Ευρώπη βρίσκεται ε, επικεφαλή σε πολύ ηγετική θέση σε ό,τι αφορά και την ευημερία των ζώων ε, και τα φυτοπαραγωγικά μέσα και το καθεξής. Όμως, αλλού βρίσκεται το ζήτημα, νομίζω. Όταν ακούω τον πρώην Επίτροπο να λέει ότι πρέπει να ε, θρέψουμε τον κόσμο για να έχουμε ειρήνη και πάλι ε, τι να πούμε για τον ε, πόλεμο με τη, Ρωσία. Ε, παραμένει λοιπόν ένα σημαντικό ζήτημα που έχει ε, επιβαρύνει πολύ τις σχέσεις μας με μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα. Το επομένω το πρόβλημα είναι αλλού. Το πρόβλημα, η κρίση που εδώ και χρόνια καταστρέφει την πλειοψηφία των ε, διαοργών μας. Και αυτή η κρίση δεν είναι τυχαία, ούτε προκύπτει από κάποια κατάρα είναι φυσική και λογική απόρρεια των ε, οικονομικών και πολιτικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θεωρώ ότι ε, εδώ και τρεις δεκαετίες όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις γνωρίζουν ότι σήμερα οι ζημίες της γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κατά τη γνώμη μου τρομερές και αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο στην αρχή δυστυχώς. Πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά γιατί είναι πολύ σημαντικά. Και πρέπει επίση ε, να συναγάγουμε συμπεράσματα, γιατί αν θέλουμε επιστημική ασφάλεια, αν θέλουμε να βελτιώσουμε την αρχή τη προφύλαξη ε, την παραγωγή, την ποιοτική, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και οι Ευρωπαίοι Γεωργοί θα έχουν τα μέσα και δυνατότητε να το πράξουν. Και όταν υπάρχει μια ε, μόνιμη αστάθεια, νομίζω ότι η βασική προτεραιότητα δεν είναι η πρόοδο, η έρευνα και η καινοτομία, αλλά να διασφαλίσουμε ένα αξιόπιστο ε, κοινωνικό και νομικό πλαίσιο για να διασφαλίσουμε την, ε, την ανεξαρτησία μας ό,τι αφορά τα επιστηστικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε κύριος Η έξπο του Μιλάνου, η Διεθνής Έκθεση του Μιλάνου και α, απηχώντα και τα σχόλια που ακούσαμε, φαίνεται ότι συνάρπασε του επισκέπτε. Σε αντίθεση με άλλε προηγούμενε διεθνεί εκθέσει, άγγιξε τον κάθε επισκέπτη, ε, τον τρόπο σκέψη του, τι παραδόσει, ε, ακόμη και τι διατροφικέ του συνήθειε. Και η Οργανωτική Επιτροπή τη ΕΞΠΟ, πολύ ορθά, διαμόρφωσε ένα πλαίσιο και νομίζω ότι αν κάτι μπορούμε να συγκρατήσουμε από την επίσκεψη στα διάφορα περίτερα της έκθεσης είναι η τεράστια ποικιλομορφία και η πληθώρα των διαφορετικών αντιδράσεων των χωρών στις διάφορες ερωτήσεις. Βέβαια, μερικά περίτερα ήταν απογοητευτικά ακόμη και μεγάλων χωρών. Αντίθετα, χώρες που υφίστανται τεράστιες δυσκολίες ε, στη γεωργία τους ε, παρουσίασαν εξαιρετικά περίπτωρα που μας έδωσαν πραγματικά ε, μαθήματα. Μας έβαλαν τα γυαλιά σε πολλές άλλες χώρες. Γιατί η διαχείριση του προβλήματος του ύδατος, ιδιαίτερα στις ε, ερημικές, στις ζώνες ε, ερήμου, δείχνουν πόσο σοβαρά είναι και τα περιβαλλοντικά μας προβλήματα και δείχνουν πόσοι χώρες αυτές, παρά την διαφορετικότητα των καθεστώτων τους, συμβάλλουν ώστε να παραμένει το γεωργικό θέμα στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Και επίσης αναδεικνύουν τη σημασία που έχει το ζήτημα της επιστηστικής ασφάλειας. Και όσοι πιστεύουν ότι είναι εύκολο και δυνατό να αγοράζουν τρόφιμα σε χαμηλότερες τιμές αλλού στον κόσμο, νομίζω ότι ένα από τα διδάγματα της επίσκεψης διαφορών, διαφορών, διαφορετικών περιπτέρων είναι ότι ακριβώς η παγκόσμια ισορροπία είναι όλο και πιο έθραυστη και θα δυσκολευτεί μεσοπρόθεσμα να θρέψει τον παγκόσμιο πληθυσμό. Και μάλιστα πήγα δύο φορές στο Μιλάνο στην ΕΞΠΟ Και μάλιστα επειδή εκλέγομαι σε γειτονική περιοχή του Μιλάνου μπόρεσα να συναντήσω και πολύ κόσμο από εκεί και βλέπω ότι αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε παγκοσμίω τον επιστηστικό κίνδυνο. Και αυτό είναι από τα σημαντικότερα διδάγματα που μπορέσαμε να αντιλήσουμε από την Παγκόσμια Έκθεση του Μιλάνου. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας να αξιοποιήσουμε αυτά τα διδάγματα και τα βιώματα εκατομμυρίων επισκεπτών αυτή τη ΕΞΠΟ που πραγματικά ήταν εξαιρετικά οργανωμένη. Και σε επισκέψεις που έκανα στην ΕΞΠΟ ακόμη και στα πλαίσια της αντιπροσωπείας, ε, δεν ε, ένιωσα ε, αρνητικές πίεση εντυπώσεις. Νομίζω ότι υπήρχε τέτοια πληθώρα διαφορετικών προτάσεων και τέτοιο πλούτος που ο καθένας μπορούσε να βρει κάτι που να τον ενδιαφέρει. Επίσης, το περίπτωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θεωρώ ότι ήταν απογοητευτικό σε σχέση με την προεργασία που έγινε και το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα γεωργικά θέματα, αλλά και σε σχέση με τη θέση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη γεωργία γενικώ και ε, δεδομένη τη μεγάλη σημασία και του ε, μεγάλου όγκου του γεωργικού προπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πετήρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμμετείχα στην παγκόσμια διάσκεψη για το Διεθνές Πρόγραμμα για την Παγκόσμια Επιστηστική και Διατροφική Ασφάλεια που έγινε στο Μιλάνο στα πλαίσια της ΕΞΠΟ. Ήμουν μέλος της επίσημης αντιπροσωπείας του πάνελ της ΤΟΑ και συμμετείχα με την κυρία Μέρη Μαγκίνε, την αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον κύριο Παύλο Ρούμπιχ, εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην παγκόσμια αυτή διάσκεψη. Τροφή για τον πλανήτη, ενέργεια για τη ζωή. Αυτό ήταν το σύνθημα της Expo του Μιλάνου και νομίζω ότι ε, είναι από τους πιο επιτακτικούς ε, στόχους και τις πιο σημαντικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πώς θα συζητήσουμε, πώς θα θρέψουμε τον πλανήτη, πώς θα εξασφαλίσουμε την επιστημιστική και διατροφική μας ασφάλεια. Αυτό είναι σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη θέση στην καινοτομία και στην έρευνα που θα συμβάλλουν ε, σημαντικά στην ε, υλοποίηση αυτού του στόχου. Το θέμα της πείνας στον κόσμο δεν είναι ζήτημα τροφίμων, αλλά θέμα πολιτικό. Και η λύση για την εξάλληψη της, ε, της πείνας δεν βρίσκεται στη γενετική τροποποίηση των προϊόντων, θα καταπολεμήσουμε, θα εξαλείψουμε την πείνα, αν κάνουμε μια ορθή και δίκαιη ανακατανομή των πόρων, του φυσικού πλούτου και των τροφίμων. Ε, γιατί κάθε χρόνο περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνους τρόφιμα σπαταλούμε και πετάμε. Και μάλιστα 100 εκατομμύρια τόνους σπαταλούμε και πετάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο. Ενώ έχουμε 850 περίπου εκατομμύρια πεινασμένου ανθρώπου ε, και αυτό ο αριθμό δυστυχώ καθημερινά μεγαλώνει και αυξάνεται. Θα πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν τι πολιτικέ μα, τον τρόπο σκέψη μα και τη μέχρι τώρα προσέγγιση μα. Και αυτό ήταν και ένα από τα αντικείμενα που μα απασχόλησαν στην έξπο του Μιλάνου. Επισκέφθηκα πολλά περίπτερα και πέραν του περιπτώρου της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης με εντυπωσίστηκε και το περίπτωρο του Βατικανού που ήταν ίσως ένα από τα πιο απλά και λιτά και απέριτα περίπτερα αλλά και από τα πιο συγκεκριμένα γιατί έδειξαν πόσο συμβάλλει η Καθολική Εκκλησία στην ε, βοήθεια των φτωχών και πεινασμένων του κόσμου και πόσο στηρίζει την οικογένεια και τον οικογενειακό πυρήνα. Και μάλιστα προσπαθεί να εξασφαλίσει την ευλογία του, του, της τροφής για όλους, γιατί δυστυχώς δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτό. Ο κύριος Αντριέ. Oui, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Φίσλερ για τα όσα μας είπε. Παρότι έφτασα καθυστερημένος ε, στην ε, συνεδρίαση, Ευχαριστώ για τα όσα έχει κάνει και ο κύριος Δεκάστρο για την διοργάνωση της έκθεσης ε, του Μιλάνου 2015. Και εγώ είχα τη δυνατότητα να παρευρεθώ και παρακολούθησα το του ε, και τη διοργάνωση και το περιεχόμενό της. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι όντως υπάρχει ένα βασικό στοιχείο που θέσατε και εσεί, κύριε Φίσλερ. Αναδείξατε ότι η επιστημική ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται ένα από τα κύρια στοιχεία της ασφάλειας στις βασικές διαστάσεις. Και σήμερα περνάμε μια, μια τέτοια δύσκολη περίοδο που μας δείχνει ακριβώς ότι αυτό είναι πραγματικό. Όλοι σχεδόν συμφωνούμε για το ζήτημα της επιστημιστικής ασφάλειας. Και το ερώτημα που τίθεται και το βλέπουμε και εμείς καθημερινά στη δουλειά μας και όπως ε, προέκυψε και από την έκθεση του Μιλάνο είναι το πώς ακριβώς θα το καταφέρουμε αυτό το στόχο που έχουμε θέσει. Για την πρόσβαση δηλαδή στην επιστημική ασφάλεια, τελικά ε, βλέπουμε δύο επιλογές. Πρέπει οι μεν να τρέφουν τους δε ή να κατευθύνουμε προς μία προσέγγιση που να προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες όλων και κατά πόσο αυτές οι δύο επιλογές είναι συμβατές μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο που πρέπει να θέσουμε σήμερα. Είναι συμβατές ή όχι. Και ανάλογα με την επιλογή που θα διαλέξουμε θα μπορέσουμε να εξελίξουμε και την έρευνα και καινοτομία. Δηλαδή, μήπως πρέπει να αναπτύξουμε την έρευνα και καινοτομία στην υπηρεσία και στο όφελο ορισμένων που μεγαλώνουν και γιγαντώνονται συνεχώς τα συμφέροντα δηλαδή των μεγάλων πολυεθνικών που θέλουν να θρέψουν υποτίθεται τον υπόλοιπο πλανήτη ή αναπτύσσουμε την έρευνα και γενοτομία για να επιτρέψουμε σε αυτούς που βρίσκονται ε, στην Ήπεθρο να τραφούν και μετά να τρέψουν και τους υπόλοιπους. Η έρευνα και η καινοτομία λοιπόν είναι βασικά στοιχεία, πολύ σημαντικά, τα βλέπουμε καθημερινά. Είναι και χωροταξικό ακόμα. Συγγνώμη, ε, το ζήτημα είναι ευρύτερο, αφορά όλους τους ε, κλάδους της επιστήμης και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το καθορίσουμε συλλογικά. Και μόνο έτσι μπορούμε να θέσουμε την έρευνα και στο όφελος ε, ε, του πληθυσμού. Βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή μία συγκέντρωση της παραγωγής ε, σε βάρος των πληθυσμών. Και θα πρέπει λοιπόν να τεθεί ο στόχος πριν αναπτύξουμε ε, τα μέσα και τα εργαλεία. Και επανέρχομαι, κλείνοντας, αυτό που είπατε κι εσείς, ναι, η γεπιστική ασφάλεια είναι πολύ σημαντική. Είναι θεμελιώδες στοιχείο ε, της ε, ασφάλειας, όμως δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο μία κινητήριο δύναμη. Να υπάρχει δηλαδή διαβούλευση με όλους τους φορείς. Και στο φορά τη τεχνογνωσία την καινοτομία πράγματι υπάρχει και τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη. Όμως το θέμα δεν είναι ο μόνος ερευνητής. Και ο ίδιος ο Γιώργος τα γνωρίζει και έχει και το συμφέρον του να τα αναπτύξει. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για να μπορέσουν όλοι να ανταλλάξουν ακόμα και τις εμπειρίες που έχουν και οι ίδιοι γεωργοί ε, στα χωράφια τους. Μάλιστα. Εξαντλήσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Όσοι είχαν ζητήσει το λόγο μπόρεσαν και μίλησαν. Οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για να απαντήσουν ή να σχολιάσουν αυτά που ακούσαμε. Δεν ξέρω με τι σειρά θέλετε να λάβετε το λόγο. Μάλλον ο γενικός ε, εντεταλμένο ε, τη συμμετοχής, για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σα και τι απόψεις σα. Νομίζω ότι μια ε, καθολική και παγκόσμια επιστημιστική ασφάλεια θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα τη ανθρωπότητας μέχρι το 2050. Αφενός αυξάνεται ο πληθυσμός, με επιστημιστικές συνήθειες και διατροφικές συνήθειες που συνεχώς αλλάζουν και άνοδο των, του βυτικού επίπεδου που επηρεάζει αυτές τις διατροφικές συνήθειες. Παράλληλα έχουμε και την κλιματική αλλαγή που συνδέεται με την έλλειψη ε, υδρία. ιδίως στα πλέον ε, φτωχά τμήματα του πλανήτη έχουμε και σοβαρή λειψιδρία και το να διασφαλίσουμε τα επόμενα χρόνια ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα από στρατηγική σκοπιά είναι από τα πλέον σημαντικά ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δραματίσει ηγετικό ρόλο σε αυτό το θέμα, όπω συνέβη και με την κλιματική αλλαγή και τη συμβολή τη ε, στην διαδικασία συμφωνία ε, των ε, στόχων αηφόρου ανάπτυξη. Είμαι πεπισμένο ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι κρίσιμο στοιχείο. Και για να γίνει αυτό πρέπει ε, να ε, συνομιλήσουμε με όλα τα ενδιαφέρουνα μέρη. Δεν αρκεί μόνο να βάζουμε σε μια αίθουσα τους επιστήμονες. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πρέπει και η ίδια κοινότητα των γεωργών, οι ίδιοι δηλαδή από όλο τον κόσμο να εμπλακούν άμεσα με, μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση και σε επιμέρους περιφέρειες ε, και φορείς από όλες τις περιοχές του κόσμου. Νομίζω ότι τα όσα έχει κάνει η Επιτροπή της οποίας προείδρευσε ο ε, Φίσλερ ήταν εξαιρετικά σημαντική. Οι Επίτροποι ε, Χόγκαν και Μόιντας συνεργάζονται πολύ στενά σε αυτό το ζήτημα και ο Επίτροπος Μόιντας ήδη ανέφερε το ζήτημα του ερευνητικού χώρου ε, διατροφής και νομίζω ότι μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα διατροφής ε, για το 2016 και μέχρι τότε θα υπάρξει μια επίσημη ανακοίνωση θεωρώ για αυτό το ζήτημα. Έχω την αίσθηση ότι το γενικότερο επίπεδο επίγνωσης ε, και ευαισθητοποίησης των ζητημάτων που άπτονται της επιστημικής ασφάλειας ήταν εξαιρετικά ε, σαφή και έτυχαν ευρεία υποστήριξη από όλου του επισκέπτε. Νομίζω ότι σε πολλά περίπτερα δόθηκε αυτή η εντύπωση. Και σημειώνω και αυτό που είπε και ο κ. Νταντάουν, ότι πραγματικά υπήρχαν πολλά εξαιρετικά περίπτερα και όχι πάντα από τις πιο πλούσιες περιοχές του κόσμου, που πραγματικά έδωσαν ένα πολύ θετικό μήνυμα ε, σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως είναι η λειψιδρία. Νομίζω ότι οι επισκέπτες που ήρθαν είτε στο ευρωπαϊκό περίπτερο είτε στα υπόλοιπα, σε γενικές γραμμές έφυγαν με ένα πολύ σοβαρό μήνυμα, ότι ο κόσμος κάτι πρέπει να κάνει. Και εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να συνεργαστούμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεργαστούν και στο μέλλον για την επίτευξη αυτών των στόχων το καλύτερο θα ήταν να δώσω το λόγο στο Franz Φίτσλερ για να απαντήσει ή να προσθέσει κάτι που θα ήθελα από πλευρά τη Επιστημονική Επιτροπή. Παρακαλώ. Πολύ ωραία. Ε, θα μου επιτρέψετε τώρα να χρησιμοποιήσω και μια άλλη γλώσσα που ξέρω. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Η Επιστημονική Διευθύνουσα Επιτροπή δεν επηρέασε επουδενή τη διαμόρφωση οποιοδήποτε περιπτέρου. Διότι εμείς ε, προσκληθήκαμε απλά και μόνο για να συζητήσουμε ένα πρόγραμμα ε, έρευνας και ανάπτυξης. Και αυτό κάναμε. Αν θέλετε δηλαδή, εμείς απλά ε, κάναμε το καθήκον μας και αυτό που μας είχαν ζητήσει δεν ήταν αν θέλετε να καταθέσουμε προτάσεις για μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής ή της γεωργικής πολιτικής της Βραζιλίας δεν μας είχαν ζητήσει κάτι τέτοιο. Και το δικό μας το καθήκον δεν ήταν επίσης να παρουσιάσουμε κάποιες ε, ιδεολογικές απόψεις στον τομέα της γεωργίας. Ξέρω ότι υπάρχει πληθώρα τέτοιων απόψεων, αλλά δεν ήταν αυτή η δική μας η δουλειά. Η δική μας η δουλειά ήταν ε, να παρουσιάσουμε γνώση και όχι απόψεις ε, και να πω και κάτι άλλο ώστε αξιότιμη κυρία να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Κοιτάξτε, Διατομεακή συνεργασία σημαίνει ότι συνδυάζονται οι διαφορετικές επιστήμες. Αυτό που δείξατε εσείς, ε, το έδειξα και εγώ και το είπα, ότι αυτό είναι πολυτομεακότητα που σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνονται πράγματι και η γεωργία και η πολιτική και η οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτές τις δύο έννοιες ε, οφείλουμε να τις χρησιμοποιούμε με σωστό τρόπο. Το ίδιο εξάλλου ισχύει και για τη συστημική, όπως αποκαλείται, σκέψη. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του παρελθόντος σε πάρα πολλούς τομείς, όχι μόνο στη γεωργία, αν δείτε ας πούμε γενικά την αναπτυξιακή πολιτική ένα πολύ μεγάλο λάθος ήταν ότι υπήρχαν παρεμβάσεις ε, στιγμιές δηλαδή αν ήθελε κάποιος να βοηθήσει μια περιοχή στην Αφρική να αναπτυχθεί δεν παίζει ρόλο μόνο η γεωργία, ε, συμπλέουν πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες και μόνο εφόσον αυτοί οι παράγοντες ε, συνδυαστούν, μόνο τότε υπάρχει η ευκαιρία πραγματικά να επιφέρει κανείς ανάπτυξη. Άρα δηλαδή αυτό σημαίνει συστημική σκέψη. Ο στόχος είναι να δεχτούμε ότι και το σύστημα των τροφίμων ανά τον κόσμο είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και οφείλουμε να μάθουμε, να, οφείλουμε να εξοικειωθούμε με αυτή την ε, πολυπλοκότητα και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι. Ίσως ε, αυτό που δεν ανέφερα στην ε, εισαγωγή, αλλά θα το πω τώρα γιατί είναι πολύ σημαντικό, πράγματι είναι αλήθεια ότι υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων που υποφέρουν από λοιμό, πείνα και κακοδιαχή και κακή διατροφή. Υπάρχουν όμως ακόμα πιο πολλοί που υποφέρουν από λάθος διατροφή. Το γεγονός ότι υπάρχει πείνα στην Αφρική οφείλεται σε μεγάλο βαθμό Εν τω μεταξύ στο ότι σε άλλες χώρες του κόσμου είμαστε αναγκασμένοι να ε, καταβάλουμε πάρα πολλά κονδύλια για να αντιμετωπιστεί το αντίθετο πρόβλημα. Η παχυσαρκία παραδείγματος χάρη. Αυτοί έχουν και αυτοί πρόβλημα και κάπως και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχω πει ότι στη Γερμανία, μόνο στη Γερμανία, ανά έτος 100 δις ευρώ δαπανώνται για να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία. Και για φανταστείτε τι σημαίνει αυτό να τον κόσμο. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα είναι τεράστιο πρόβλημα στις ε, αναδυόμενες χώρες. Το ποσοστό των σαρκών αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο έντονο από οπουδήποτε αλλού στο Μεξικό. Άρα δηλαδή και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όσον αφορά τώρα το ρόλο της Ευρώπης το νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Διότι εγώ δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Δεν είναι αλήθεια ότι το καθήκον της Ευρώπης είναι να προσφέρει επισητιστική επάρκεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Όχι, εμείς οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε ή δυνατόν τα περισσότερα τρόφιμα να παράγονται και να τίθενται σε εμπορία επιτόπου όχι να μεταφέρονται τα τρόφιμα ανά τον κόσμο. Αυτή δεν είναι καλή στρατηγική. Και είναι αλήθεια ότι σε εμά στην Ευρώπη ο γεωργικός τομέας αυτή τη στιγμή δεν είναι παντού αηφόρος. Εντατικοποίηση της αηφορίας, αυτή είναι μια έννοια που χρησιμοποίησε πριν από κάποια χρόνια η Βρετανική κυβέρνηση εντατικοποίηση της αηφορίας σημαίνει όχι να αυξηθεί παντού η παραγωγή αλλά σημαίνει σε κάποιους τόπους και σε κάποια συστήματα να ασχοληθεί κανείς περισσότερο με το περιβάλλον και όχι με την παραγωγή τροφίμων. Αυτά πρέπει κανείς να έχει κατά νου αν θέλει να προχωρήσει. Πρέπει λοιπόν να σας πω, τελειώνοντας, αν θα μπορούσα να εκφράσω μία παράκληση ή μία επιθυμία, γιατί αυτό ήταν και μία μεγάλη επιθυμία, μία ουσιαστική επιθυμία των επιστημών που συμμετείχαν στις συζητήσεις μας. Δεν πρέπει να πιστεύετε ότι σήμερα στην Ευρώπη, τουλάχιστον όσον αφορά την έρευνα στη γεωργία, είμαστε στην πρώτη θέση ανά τον κόσμο. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ε, δέστε λιγάκι ε, χώρες όπου η Βραζιλία και όλο και περισσότερο η Κίνα ε, αυτά τα θέματα της γεωργικής έρευνας ερευνώνται πολύ πιο συστηματικά και εκεί δαπανώνται πολλά περισσότερα κονδύλια στη γεωργική έρευνα από ό,τι σε εμά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα και εγώ να σας παρακαλέσω να το ελέγξετε λιγάκι αυτό στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές όσον αφορά τις δαπάνες για, τα, την έρευνα. Έχει προσημειωθεί ένα κονδύλι για τις γεωργικές έρευνες και για δέστε λιγάκι ε, ποιο είναι το κονδύλι αυτό και τότε θα μπορείτε να δείτε κατά πόσον τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν είναι τα σωστά ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι η κοινωνία πρέπει να συμμετέχει στην πολιτική έρευνα και πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη συμμετοχή των πολιτών. Κατά τα άλλα, και αυτό είναι μία παράκληση εκ μέρους μου, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι η Ευρώπη να παραμείνει στην κορυφή οποτεδήποτε γίνεται λόγος για την παγκόσμια επισητιστική ασφάλεια. Και το μόνο που μπορεί να μας ενδιαφέρει είναι αυτή η παγκόσμια επισητιστική ασφάλεια. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο δεν είναι δυνατόν αυτή την ε, ασφάλεια να την κατακαιρματίσει. Και το γεγονός ότι πρέπει να παρεμβαίνει κανείς καθοδηγητικά, αυτό είναι σωστό. Αλλά και το ότι πρέπει να παρεμβαίνει σωστά, νομίζω αυτό πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Γιατί δεν υπάρχει μία εφάπαξ κίνηση και μετά τίποτα άλλο. Πρόκειται για μια εντολή που θα μας συνοδεύει όλους μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως επίσης και η εντολή την ε, γεωργική πολιτική να την μεταρρυθμίσουμε με συγκεκριμένα βήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα ήθελα να σας προσκαλέσω, να σας καλέσω να δείτε λιγάκι αυτό το ενημερωτικό δελτίο για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως και εκεί θα δείτε ότι τόσο το θέμα των εισαγωγών το οποίο το δείξατε και πολύ σωστά ε, περιλαμβάνεται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο αλλά και πολλά άλλα ε, ερευνητικά θέματα και δεν είναι δυνατόν σε πέντε λεπτά όλα αυτά να τα εντάξει κανείς σε μια εισήγησή Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Νομίζω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το στοιχείο για τα 800 εκατομμύρια ανθρώπους ε, που έχουν πολύ δύσκολη πρόσβαση στη, στα στην τροφή, στα τρόφιμα. Δεν είναι όλα αυτά τα 800 εκατομμύρια άνθρωποι που λιμοκτονούν, που πεινάνε, αλλά που ίσως υποσυτίζονται ή δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα τρόφιμα. Πάντως πολύ σωστά είπε ο κύριος Φίσλερ ότι θα αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις γνώσεις και τις εμπειρίες που συγκεντρώσαμε για τις ε, προτάσεις που θα κάνουμε για την κοινή γεωρική πολιτική και στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία, ο Επίτροπος Χόγκαν διοργάνωσε ε, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Καινοτομία και Έρευνα πολύ σημαντική διάσκεψη στην οποία αναφέρθηκαν όλα αυτά τα συστήματα. Και τον Απρίλιο ή τον Μάιο θα υποβληθεί και η, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το ρόλο της καινοτομία και της έρευνας στη γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως ε, που συνέβαλε τα μάλα στην ε, διοργάνωση της αντιπροσωπείας μας για την έξπο του Μιλάνου και έκανε γενικώ πολλές προσπάθειες ε, για τη συμμετοχή μας εκεί. Και να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας, τον κύριο Βίλκινσον και τον κύριο Φίσλερ που ήρθαν, μας παρουσίασαν τις ε, απόψεις τους, τα απορίσματα των ομάδων τους ε, και ο κύριος Φίσλερ μάλιστα μας παρουσίασε και το εγχειρίδιο αυτό, το ενημερωτικό βιβλιάριο για την Expo. Ήταν πολύ σημαντικές νομίζω ε, οι εργασίες που έγιναν στα πλαίσια αυτής της πολύ σημαντικής οργάνωσης, της ΕΞΠΟ του 2015 και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν και συμμετείχαν ε, στην προσπάθεια αυτή και πρώτα απ' όλα στον Πρόεδρό μας τον κύριο Δεκάστρο. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι θερμά τους καλεσμένους μας και ένα σύντομο διάλειμμα δίλεπτο για να τους ξεπροβοδίσουμε. na Περιμένουμε πάντως τις επόμενες πρωτοβουλίες και από εσάς και την Επιτροπή. Państwa, przechodzimy. Bardzo Σας ευχαριστώ λοιπόν συνάδελφοι για τη συμμετοχή στη συζήτηση του σημείου 4. Περνάμε στο σημείο 5 τώρα με θέμα την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Τροποποίηση του κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ε, που αφορά τους επίσημους ελέγχους και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου. Ο εισηγητής μας για το θέμα αυτό είναι ο κύριος Χόισλινγκ. Θα μας ενημερώσει για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου έγιναν μέχρι στιγμής τρεις τέτοιοι τριμερείς διάλογοι, δύο επί Λουξεμβουργιανής και ε, Ολλανδικής Προεδρίας, ο τρίτος τριμερείς διάλογος ε, επίκειται στις 29 Φεβρουαρίου. Οι διαπραγματεύσει είναι δύσκολε από πολιτική άποψη και περίπλοκε από τεχνική άποψη. Ο εισηγητή μα είπε ότι είναι ο κύριο Χόισλινγκ, που είναι και ο κατάλληλο να μα ενημερώσει για το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και δύσκολο το θέμα της βιολογικής γεωργίας και της επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων και είναι δύσκολο και από πολιτική αλλά και περίπλοκο από τεχνική άποψη, όπως σας είπα. Και μετά θα δώσουμε το λόγο και σε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά είπατε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο θέμα. Οι διαπραγματεύσει δεν είναι απλές. Ε, μέχρι τώρα είχαμε τρεις ε, τριμερείς ε, διαλόγους, δύο υπό την Προεδρία του Λουξεμβούργου θα θέλαμε να έχουμε και άλλους, και άλλες τέτοιου είδους συζητήσεις, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά προς το τέλος μια Προεδρία εστιάζει την προσοχή της σε θέματα που θέλει να κλείσει. Ε, τώρα, με την νέα Προεδρία είχαμε ήδη μία και στις 29 έχουμε τη δεύτερη τριμερή συνάντηση. Μέχρι τον Ιούνιο θα ακολουθήσουν έξι περαιτέρω τριμερείς συζητήσεις. Τώρα, κατά πόσο θα κλείσει το θέμα, η Προεδρία βέβαια, η νυν Προεδρία, έχει πει ότι ενδιαφέρεται διακαώς ε, να συμφωνήσουμε, αλλά υπάρχουν πολλά θέματα που είναι ακόμα ανοιχτά, θα σας τα εξηγήσω. Και πρέπει να υπογραμμίσω ότι η κατάσταση στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλή. Ε, σε πάρα πολλά θέματα προχωράμε. Ε, είχαμε και πολλές ε, τεχνικές αντίσεις όπου προσπαθήσαμε να επιτύχουμε συμβασμούς. Όπως είπε λοιπόν και ο Πρόεδρος, σημειώνουμε κάποια πρόεδρο όμως, ξέρετε κάτι, δεν πρέπει τελικά όλα αυτά να είναι εις βάρος της ποιότητας. Το λέω αυτό ξεκάθαρα, γιατί ε, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ε, κάτι τέτοιο ούτε στους γεωργού ούτε στους εμπόρους. Λάθη που δεν θα μπορούμε να διορθώσουμε. Υπάρχουν άρθρα δύο-1, μιλήσαμε για το πεδίο εφαρμογής, μιλήσαμε για τους ε, ορισμούς, για τις διατάξεις παραγωγής και στην τελευταία στον τελευταίο τριμερή διάλογο ασχοληθήκαμε ουσιαστικά με το θέμα των εισαγωγών. Αυτός είναι ένας ε, τομέας όπου ε, θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε το των δυνατών, όμως λεπτομέρειες είναι δύσκολες. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή, ε, πρέπει να εξηγήσουμε ποια προϊόντα θα συμπεριληφθούν στη συμφωνία και ποια όχι. Στο παράρτημα συμφωνήσαμε ότι η Κομισιόν θα προσθέσει προϊόντα που διέπονται από καθεστώς ε, κατεξοδότηση πράξεων. Πάντως, πάνω σε αυτό δεν έχουμε καταλήξει και το Κοινοβούλιο μου έχει δώσει την εντολή να συμπεριλάβουμε και το θέμα της ε, κοινοτικής σύντησης ε, στον κανονισμό και δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα στο θέμα των ε, φυτών, του φυτικού υλικού, ε, των ε, φυτών που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτική χρήση. Όσον αφορά τους στόχους και τις αρχές, πολλοί μπορεί αυτά να μην τα βρίσκουν σημαντικά, αλλά έχουν ασκούν επιρροή στη νομοθεσία. Στόχοι και αρχές λοιπόν δεν διαφοροποιήθηκαν στην προηγούμενη πρόταση της Επιτροπής. Τελικά όμως συμφωνήσαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός και παραδείγματος χάρη στους στόχους πρέπει να διευκρινίσουμε ε, κατά πόσον ε, τα τοξικής, ε, τα τοξικά προϊόντα επηρεάζουν τον άνθρωπο. Αυτά είναι έτσι κάπως γενική φύσεως θέματα, τα οποία πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε έτσι να μην υπάρχουν ασάφειες. Εκεί που δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα και αυτό είναι σημαντικό, ε, γνωρίζω ότι οι συνάδελφοι από τις ε, βόρειες χώρες ανησυχούν πάρα πολύ γι' αυτό, το εξή. Σε ποιο βαθμό η γεωργία, η βιολογική γεωργία πρέπει να δεσμεύεται να είναι μόνο ε, στο έδαφος. Έχει τεθεί το θέμα των ε, θερμοκηπίων. Πάντως για τις βόρειες ε, περιοχές πρέπει να βρούμε κάποια λύση, να μην προχωρήσουμε πάρα πολύ, γιατί σε αυτές τις χώρες υπάρχει βιολογική παραγωγή στα θερμοκήπια και αυτή πρέπει να μπορεί να συνεχιστεί. Επίσης έγινε συζήτηση για τις μικτές επιχειρήσεις. Αυτό αντιμετωπίζεται με διαφορετικούς τρόπους στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε καταρχήν όχι μεικτές επιχειρήσεις. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν διαφορετική άποψη από αυτού. Όμως και εμείς καταστήσαμε απόλυτα σαφές, σημαντικό αυτό, ότι στο μέλλον θα υπάρχουν μεικτές επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να ε, διαχωριστούν ξεκάθαρα οι μονάδες παραγωγής. Δεν είναι δηλαδή στην ίδια επιχείρηση να υπάρχουν ε, ε, βιολογικές αγελάδες μαζί με άλλες μη βιολογικές που εκτρέφονται δηλαδή με μη βιολογικό τρόπο. Ε, αυτό ο καταναλωτής, το διαχωρισμό τον βρίσκει σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν σαφής διαχωρισμός των παραγωγικών μονάδων και εγκαταστάσεων μέσα σε μια επιχείρηση, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα των ε, βιολογικών ζωοτροφών. Η αλλαγή κάποιες επιχείρησης το να γίνει βιολογική δεν πρέπει να δυσχεραίνεται. Έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο να περάσει κανείς από την παραδοχησιακή στη βιολογική γεωργία. Δεν χρειάζεται να το κάνει πιο δύσκολο. Τώρα, ε, απαγόρευση των ε, ε, γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων. Προφανώς και δεν επιτρέπονται αυτά στη βιολογική γεωργία, θα το εξηγήσει ο συνάδελφος. Και στις εισαγωγές θα πρέπει να προσέχουμε έτσι ώστε όπου δεν, ισχύ, όπου δεν υπάρχουν κανονισμοί για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ε, στις χώρες προέλευσης να ισχύουν αυτοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω επισημάνει το τι πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Σας είπα κατά κύριο λόγο ο κανονισμός για τις εισαγωγές. Ως κοινοβούλιο είπαμε ότι χρειαζόμαστε ένα σαφή κανονισμό να ισχύει η συμμόρφωση, δηλαδή οι εισαγωγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσαρμόζονται και συμμορφώνονται στην κείμενη νομοθεσία. Αυτό μπορεί να ισχύει σαν αυτονόητο, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Ε, χρειαζόμαστε και κανόνες ε, συμμόρφωσης οι οποίοι πρέπει να θεσπιστούν να μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι θα βρούμε κανόνες με βάση τους οποίους όταν εισάγεται κάτι από τρίτες χώρες με τις οποίες δεν έχουμε συμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να συνάψει συμφωνίες. Αυτό δεν θα είναι εύκολο για πολλές χώρες. Ο στόχος και του Συμβουλίου και της Επιτροπής είναι να περιοριστεί ο αριθμός των εξαιρέσεων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι απλό στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή ε, το πώς μπορούμε ναι με να απλωστεύσουμε τους ελέγχους αλλά να μην ε, θέσουμε σε κίνδυνο την τήρηση των ε, προδιαγραφών και να μην υπάρξουν εξαιρέσεις στις προδιαγραφές. Επ' αυτού μπορούμε να επανέλθουμε στον επόμενο τριμερή διάλογο. Οι τεχνικές ομάδες ήδη ασχολούνται με τις ε, προκατακτικές εργασίες για να καταλήξουμε σε κανονισμό συμφωνία. Σας λέω, με απόλυτη, με απόλυτη, σας λέω κατηγορηματικά ότι αν καταλήξουμε τελικά αυτό δεν θα γίνει εις βάρος της ποιότητας. Οι βιολογικές καλλιέργειες είναι υψηλού επίπεδου και δεν θέλουμε να ε, θεσπίσουμε γρήγορα κανονισμούς που θα οδηγήσουν σε επιδείνωση της ε, ποιότητας. Ε, στους και ηγητές θέλω να απευθύνω τις ευχαριστίες μου. Είμαστε μια πολύ αρμονική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλω να ευχαριστήσω θερμά ε, και τη γραμματεία. Χωρίς ε, τις προετοιμασίες από την γραμματεία, κυρίως για, τις ε, τριμερείς, για τους τριμερείς δεν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τίποτα. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, αλλά είμαι σίγουρος ότι με την υποστήριξη και των άλλων ομάδων ε, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αίσιο τέλος. Αν αυτό θα είναι στις 36 θα δούμε σε τελική ανάλυση, εξαρτάται και από το κατά πόσο είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν σε συμβασμούς οι υπόλοιποι θεσμοί. Και εμείς το ίδιο σας ευχόμαστε καλή τύχη και καλή επιτυχία κύριε Χόισλινγκ. Το λόγο έχει κύριο Στάκουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημαντικά σημεία, σε δύο πολύ κρίσιμα σημεία. Και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Χόισλινγκ να τα λάβει υπόψη στην διατύπωση τη θέση του στην τριμερή διάλογο για την βιολογική γεωργία. Καταρχήν ό,τι αφορά τα θερμοκήπια. Προσοχή στην τροπολογία 276 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί προτείνουμε μόνο παραγωγή στο έδαφος, παραγωγή προϊόντος στο έδαφος, στο χώμα. Ε, ενώ το ισχύον κείμενο ε, προβλέπει land-based production και όχι soil-based, στη γη και όχι στο χώμα. Κάτι τέτοιο, αν εγκριθεί η νέα η τροπολογία αυτή, θα αχρηστευτεί η βιολογική ε, καλλιέργεια σε πολλές παραγωγές. Γιατί στη Φιλανδία, ε, επειδή έχουμε παγωνιά, δεν μπορούν ε, οι ρίζες να βρίσκονται στο έδαφος, γιατί το έδαφος είναι παγωμένο. Οπότε δεν συμφωνώ με την τροπολογία 276, είναι απαράδεκτο και νομίζω ότι αντιβαίνει στους στόχους ε, της ε, αναθεώρησης του κανονισμού. Θα πρέπει διάφοροι ε, τρόποι βιολογικής παραγωγής να συνεχίζονται στα κρατημέλη ανάλογα με τις καιρικέ τους συνθήκες. Γιατί θα πρέπει να σεβαστούμε τις εθνικές παραδόσεις και να αποφύγουμε και απώλεια της θρεπτικής αξίας των ε, βιολογικών προϊόντων. Επίσης, ο προσανατολισμός ε, στον κίνδυνο συνάδει με τους στόχους ε, της αναδιατύπωσης. Η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου είναι μια ισορροπημένη συμβαστική λύση. Και επιτρέψει τα κράτη-μέλη, εφόσον το επιθυμούν, να μειώσουν το γραφειοκρατικό άχθος για ε, παρόχους ε, που προσφέρουν χαμηλό κίνδυνο και έχουν στοχευμένους ελέγχους για ενέργειες με υψηλότερο βαθμό κινδύνου και επίσης αξιοποιούν καλύτερα τα κρατικά κονδύλια και τα κοινοτικά κονδύλια. Συμφωνούμε λοιπόν περισσότερο με την προσέγγιση του Συμβουλίου στο σημείο αυτό. Ερωτώ τον κύριο Χόισλινγκ. Πώς θα προωθήσετε αυτά τα δύο σημεία που είναι κρίσιμα και τι θέση θα λάβετε ως εισηγητής της Επιτροπής Γεωργίας στον τριμερή διάλογο που στόχο έχει την επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άγνιου παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή τη φορά ήρθε κάποιος από μια σκανδιναβική χώρα εδώ, ο μιλητή, ε, ο προλαλής σας, ε, ανέδειξε τα ζητήματα που και εγώ επισημαίνω από την πλευρά των συναδέλφων μου στη Σουηδία. Άκουσα τον Μάρτιν Χάουσλινγκ, τον κύριο Σιγητή, που συμμετείχε στην τριμερή διάλογο. Είπε λοιπόν ότι αυτό το soil link δεν έχει επιληθεί το ζήτημα του εδάφου. Όμω, Μάρτιν, ποια είναι η γνώμη σου, η προσωπική σου άποψη. Θεωρείς ότι οι Σκανδιναβοί γεωργοί θα πρέπει να λάβουν αυτή την εξαίρεση ή πραγματικά θε να επιμείνει ε, στην καθαρότερη μορφή και αυστηρότερη μορφή βιολογικής καλλιέργειας. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου προσωπική γνώμη, γιατί νομίζω ότι αυτό θα κάνει διαφορά. Είναι η Κομισιόν που το οθεί και το πιέζει ή εσύ. Μάλιστα αυτό που ανέφερες για τις ε, ανάμεικτες καλλιέργειες και εκμεταλλεύσει μάλλον, γιατί και εμείς έχουμε μεγάλες εκμεταλλεύσει στον Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορούμε να διατρέξουμε λοιπόν αυτό το ρίσκο. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει ανάμειξη ε, των ε, ζώων. Επομένω, ε, κάποια φορά συμφωνούμε κιόλας. Ανέφερε στο όνομά μου στη φορά του γενετικώ τροποποιημένου ε, οργανισμού. Αν οι πελάτε που θέλουν ε, βιολογικά δεν θέλουν να καταναλώσουν τίποτα που έρχεται σε επαφή με γενετικώ τροποποιημένου, είτε είναι ζωοτροφέ είτε καλλιέργειε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ο καταναλωτή έχει πάντα δίκιο και θα πληρώσουν παραπάνω για να το αποκτήσουν. Αυτό που εμένα με απασχολεί και ξέρω, θα ήθελα μάλλον να μου πεις αν αυτό έχει ενταχθεί στην νομοθεσία όπως θέλαμε, είναι ότι οι ε, καλλιεργητές, γεωργοί των βιολογικών μπορούν να επιβάλλουν τον τρόπο που θα καλλιεργούν οι υπόλοιποι. Δηλαδή να πούνε οι περιβαλλοντικοί φορεί ότι όχι, αν ο ένα ε, βιολογική καλλιέργεια ε, έχει την εκμετάλλευσή του εκεί, δεν μπορεί να πάει κάποιο δίπλα του και να ε, καλλιεργήσει με μεταλλαγμένα. σω μπορούσε να μα το διευκρινίσει αυτό. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Εράν Γκαρσία. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που καταλήξετε σε συμφωνία για ένα τόσο σημαντικό θέμα, αυτό των ανάμεικτων εκμεταλλεύσεων. Και στην πατρίδα μου, κυρία Άγγινιο, έχουμε το πρόβλημα αυτό των ε, μεικτών εκμεταλλεύσεων. Και αν δεν είχε βρεθεί λύση, θα είχαμε πρόβλημα με τη βιολογική παραγωγή. Γιατί η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερο παραγωγό βιολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ήταν καλή η συμφωνία στην οποία κατέληξαν Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Βέβαια, στα πολιτικά θέματα δεν έχουμε και εντυπωσιακή πρόοδο. Πολύ καιρό ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, με την βιολογική γεωργία και την επισήμεση των βιολογικών προϊόντων και ακόμη πόρο απέχουμε από τη λύση. Σας εύχομαι πραγματικά καλή τύχη και μακάρι να εποδοθεί αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό το καθεστώς στον εισαγωγό, για παράδειγμα, γιατί αν θέλουμε όντως ο Ευρωπαίος καταναλωτής να έχει εμπιστοσύνη στα βιολογικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά και εγώ είμαι η πρώτη που θα ήθελα να πολλούνται τα βιολογικά προϊόντα, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πολλούνται ισπανικά προϊόντα, μια και η Ισπανία, είναι η μεγαλύτερη παραγωγό βιολογικών προϊόντων. Θα ήθελα όμω για να ε, κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου καταναλωτή να είμαστε πολύ αυστηροί με τα τρόφιμα που περνάνε τα σύνορά μα. Ή δε θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Ε, έλλειψης ασφάλειας επισητιστικής. Και το απέχομαι εννοείται, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην δημιουργήσουμε μια επισητιστική ανασφάλεια σε ό,τι αφορά τη βιολογική παραγωγή και κλονίσουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, ιδιαίτερα σε περίπτωση εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί και να προσέξουμε τη συμφωνία θα δεχτούμε στο θέμα αυτό. Γιατί, επαναλαμβάνω, για μένα το ζητούμενο είναι να έχουμε ασφαλή βιολογική παραγωγή στην Ευρώπη και να πολλούνται όσο περισσότερα βιολογικά προϊόντα γίνεται. Ευχαριστώ κύριε Σουαζόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο καταναλωτής ε, όντως ε, ζητάει καλύτερες πληροφορίες, καλύτερη ενημέρωση. Εάν υπάρχουν μέτρα με πιο αυστηρές ε, προδιαγραφές και μέτρα, δυστυχώς ε, φοβάμαι ότι το σχέδιό μας μπορεί ε, να ευνοεί μόνο τα βιομηχανικά βιολογικά προϊόντα. Και αυτό πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει για το καταναλωτή, γιατί και για τους καλλιεργητές που μένουν εκτός αγοράς ε, ιδίω ό,τι αφορά τους μικροκαλλιεργητές που δεν μπορούν να, ε, να ανταγωνιστούν στα βιολογικά ε, και προσιτά προϊόντα τις μεγάλες πολυεθνικές. Είναι αδύνατο λοιπόν γιατί και το κάθε ε, προϊόν έχει συγκεκριμένε προδιαγραφέ και δυσκολίε χαρακτηριστικά. Ανάλογα λοιπόν και με το οικονομικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την το ελεύθερο εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα. Και πάλι μπορούν λοιπόν να διακινδυνεύσουμε τη θέση των βιολογικών προϊόντων. Επομένω, πρέπει να εξετάσουμε ε, την επιστημική ασφάλεια, τι δυσκολίε που υπάρχουν στην καλλιέργεια, τα χημικά προϊόντα και πώ αυτά χρησιμοποιούνται και το καθεξής ίσως θα πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένα πρότυπα. Ξέρουμε ότι το 100% των βιολογικών προϊόντων ε, και ε, λαχανικών εισάγονται ε, στην Γαλλία και γι' αυτό πρέπει να δούμε και το κόστος των αερίων του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής. Είναι πολύ υψηλότερη τιμή, πολύ υψηλότερη ρήπανση που προκαλείται σε σχέση με τα ντόπια προϊόντα. Για παράδειγμα, η Μπιονέστη ισπανική πολυεθνική που ε, εξειδικεύεται στις ε, ε, φράουλε, κατηγορήθηκε για κοινωνικό dumping για να ρίξει τις τιμέ. Και αναφέρουμε ότι όσο μεγαλώνει η, η απόσταση πρέπει να διανύσει κανείς για να μεταφέρει το προϊόν, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος. Επομένως, πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια και παίρνω το λόγο αμέσω μετά τον κύριο Λοζό. Θα ήθελα να εξάρω το έργο του κλάδου ε, καλλιέργειας φράουλα στη Γουέλβα. Είναι πολύ σοβαρό το έργο, ε, αξιοσέβαστο και σε καμία περίπτωση δεν κάνει ε, κοινωνικό ντάμπινγκ. Νομίζω ότι πρέπει να αναδείξουμε το έργο των ανθρώπων αυτών και των επιχειρήσεων αυτών. Νομίζω ότι είναι ανεδαφικές και αβάσιμες οι κατηγορίες που εκτόξευσε εις βάρος των ε, φραουλοκαλλιεργητών της Ισπανίας ο κύριος Λόζο. Κύριε Χόισλινγκ, θα είχατε την καλοσύνη να μου διευκρινίσετε το θέμα των εισαγωγών, γιατί συμφωνώ με την κυρία Εράνς ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το ρυθμίσουμε. Είναι προς το συμφέρον μας ε, να ρυθμίσουμε όλο το ζήτημα των εισαγωγών των βιολογικών προϊόντων. Και για τον καταναλωτή, αλλά και για τους ε, Ευρωπαίους βιολογικούς ε, γεωργούς. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε πολύ απαιτητικοί με τους δικούς μας γεωργούς ε, βιολογικής παραγωγής ε, ενώ να είμαστε πιο χαλαροί και επικείς με τα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα. Γιατί αυτό είναι άδικο εις βάρος των Ευρωπαίων γεωργών. Επίσης, αν κατάλαβα καλά κύριε Χόισλινγκ, θα προσπαθήσετε να διεκπαιρεώσετε τις εργασίες μέχρι τον Ιούνιο και να συμφωνήσετε με το Συμβούλιο. Από ό,τι ξέρω όμως, ε, πολλές είναι οι εκκρεμότητες ακόμη. Βέβαια είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν ε, οι διαπραγματεύσεις, αλλά όχι εις βάρος της ποιότητάς τους. Όχι ταχύτητα εις βάρος της ποιότητας. Αλλά ακόμη πολλής χρόνος ε, μένει, που σημαίνει ότι πολλά σημαντικά θέματα παραμένουν εκκρεμή. Επίσης, σε ό,τι αφορά την ε, ε, μεταφορά ε, γενετικών τροπημένων οργανισμών ή τη διασταυρωμένη μόλυνση, νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει λυθεί πια στις διαπραγματεύσεις. Ισχύει αυτό. Ευχαριστώ κύριο Σαντριέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά και κάπως περίεργη. Έχω την αίσθηση ότι είναι η πρώτη φορά που μιλούμε για την έκθεση αυτή για τη βιολογική παραγωγή. Ενώ την έχουμε υπερψηφίσει στην Επιτροπή Γεωργίας. Και σήμερα ε, το έργο και η αποστολή του εισηγητού μας και των σχεδόν εισηγητών είναι να προασπίσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανήκω και εγώ στους και ηγητές. Δεν θα επαναλάβουμε εδώ την συζήτηση επί της ουσίας. Αν κάθε φορά και σε κάθε στάδιο της διαπραγμάτευσης ο καθένας προσπαθεί να επαναφέρει το ζήτημα σε επίπεδο ουσίας, νομίζω δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Ούτε εξυπηρετούμε εδώ τους στόχους μας, που είναι να προωθήσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνεργασία ήταν πολύ καλή και σίγουρα θα πρέπει να επιταχύνουμε ε, τις προσπάσεις για τα τέσσερα εκρεμή σημαντικά σημεία από πολιτική άποψη. Γιατί έχουμε προχωρήσει σε θέματα τεχνικά, αλλά όχι σε θέματα πολιτικά. Το θέμα των των εκμεταλλεύσεων, για παράδειγμα. Εκεί υπάρχει όλο και μεγαλύτερη σύγκληση με το Συμβούλιο. Επίση, το θέμα των ελέγχων. Το σκεγγραφήσαμε στον τελευταίο τριμερή διάλογο, αλλά δεν οριστικοποιήθηκε η απόφαση για τους ελέγχους. Επίσης το θέμα των εισαγωγών. Και παρόλο που είναι πολύ σημαντικός ε, ο τομέας αυτός, δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για τις εισαγωγές. Και το θέμα των κατοφλίων, όπως είπε η κυρία Γκαρσία. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Κρίσιμα σημεία του νέου κανονισμού. Και υπάρχουν λοιπόν πολιτικά θέματα, αλλά και πολλά διακυβευόμενα. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τις συζητήσεις. Αλλά προσοχή, γιατί εμείς το κείμενο το συζητήσαμε, διεξοδικά το τροποποίησαμε και είναι σήμερα διαμορφωμένη και ξεκάθαρη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτή προωθούμε στον τριμερή διάλογο. Υπάρχει, όπω είπα, όλο και μεγαλύτερη σύγκληση με το Συμβούλιο. Γι' αυτό και καλό θα ήταν να επιταχύνουμε τι εργασίε, ώστε να αναδείξουμε ως προτεραιότητα ζητήματα τα πολιτικά και να τα διεκπαιρεώσουμε το συντομότερο δυνατό. Άλλωστε, πρόκειται για ένα ιδιάζοντα τομέα, για τον οποίο ήδη ισχύει κανονισμός. Εδώ μιλούμε για τροποποίηση απλώς κανονισμού, για αναθεώρηση κανονισμού. Οπότε ας πέψουμε βραδέως. Είναι επιτακτικό το θέμα, αλλά όλα είναι σχετικά. Γι' αυτό να μην βιαστούμε, για να μην σκοντάψουμε. Είναι σημαντικό να τροποποιήσουμε τον κανονισμό, αλλά να καταλήξουμε σε ένα ποιοτικό κανονισμό. Επίσης, ο νέος κανονισμός για τη βιολογική γεωργία δεν θα πρέπει να, να διεκπαιρεωθεί άρων-άρων, γιατί αφορά πολύ σημαντικά θέματα και νομίζω ότι είναι καθήκον και ευθύνη μας να είμαστε πολύ ακριβείς στην έκβαση του τριμερούς διαλόγου, τα αποτελέσματα του οποίου θα σας τα παρουσιάσουμε διεξοδικά. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μαγιόλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε προλαλή σα, Δηλαδή έχουμε προχωρήσει αρκετά σε αυτά που είχαμε συμφωνήσει στο Κοινοβουλίο και ενώ ώψη αυτό έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η μία φορά κάτι που λέγεται προηγουμένως σχετικά με τους ελέγχους. Ο κύριος τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την, ε, το δυναμισμό που δείχνει στους ε, τριμερείς ε, διαλόγους. Για τους ελέγχους όμως δεν είπε τίποτα και νομίζω ότι το είχαμε συμφωνήσει αυτό. Δηλαδή θέλουμε να διατηρήσουμε τους ετήσιους ελέγχους και πάντα με, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση κινδύνου. Αν όμως ακολουθήσουμε μόνο το δεύτερο σκέλος, την αξιολόγηση κινδύνου, ε, δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να συνεχιστούν και οι κανονικοί έλεγχοι. Δεύτερο, σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ο κύριος ε, Χόισλινγκ είπε ότι οι οργανισμοί αυτοί δεν επιτρέπονται, απαγορεύονται στις οικολογικές καλλιέργειες. Όμως βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συζήτηση. Δηλαδή, τι είναι τελικά γενετικά τροποποιημένο, αυτό πρέπει να το απαντήσει η Κομισιόν. Οι τελευταίες ε, διαδικασίες όπου στο τελικό προϊόν δεν μπορεί κανείς καν να ελέγξει αν έχουν εντωμεταξύ χρησιμοποιηθεί γενετικά τροπημένοι οργανισμοί στην αλυσίδα παραγωγής ή όχι. Αυτό θέλω να ξέρω αν το συζητήσετε στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη ικανοποίηση ότι υπάρχει εξέλιξη και πρόοδος ό,τι αφορά τις ε, ε, μοιρασμένες αυτές μικρές Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να επιτρέψουμε ε, μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας ε, και τους επιτρέπει να μπουν ε, σταδιακά σε αυτή τη νέα τεχνολογία. Τώρα, με λύπη ακούω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι από τη Βόρεια Ευρώπη. Θα ήθελα το σύνολο της Ευρώπης ε, να ε, πάρει μια κοινή θέση σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα και ότι συμβαίνει με τις ε, καλλιέργειες εκτός εδάφους που μπορούν να γίνουν σε θερμοκήπια. Έτσι, χάνουμε την εικόνα αυτή την αρχική των βιολογικών προϊόντων και χάνουμε και τον τελικό μας σκοπό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των εισαγωγών. Θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα το οποίο ελπίζω να βοηθήσει και ε, στην διαπραγμάτευση. Σταδιακά προχωρήσαμε στην απαγόρευση της χρήσης ορισμένων προϊόντων ε, και εναέριων ε, στεκασμών σε συγκεκριμένες γαλλικές περιοχές. Τα ελικόπτερα αυτά και τα αεροσκάφη τα έχει αγοράσει η Δομινικανή Δημοκρατία και σήμερα αυτός ο εξοπλισμός βοηθάει ε, στην ε, εκμετάλλευση που αφορά την ε, μπανάνα σε αυτή τη χώρα. Επομένως, πρέπει να είμαστε όντως πολύ προσεκτικοί στη διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά το κριτήριο της αμοιβαιότητας. Γνωρίζω ότι οι συνέδελφοι από το Διεθνές Εμπόριο έχουν διαφορετική γνώμη από αυτούν. Η αμοιβαιότητα συνήθως τη βάζουμε παντού σε ό,τι αφορά το δικό μας ε, θέμα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θέλουμε στους Ευρωπαίους πολίτες να πουλάμε προϊόντα εισαγωγής που όμως να ξεπερνούν τους κανόνες που ε, ισχύουν σε συγκεκριμένους δικούς μας ευρωπαϊκούς τομείς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε τον Μαρτίν ε, για την ανασχόλησή του με αυτό το δύσκολο θέμα. Οι βιολογικές ε, καλλιέργειες καλά τα πήγαν μέχρι τώρα με τον σχετικό κανονισμό και εγώ πιστεύω ότι όσον αφορά τον νέο κανονισμό δεν πρέπει να βιαστούμε, δεν πρέπει να εμποδίζουμε τις βιολογικές ε, καλλιέργειες. Κάθε άλλο Πρέπει να φροντίζουμε να τηρούνται οι προδιαγραφές και στις αγωγές και στην ίδια παραγωγή ε, και κάτι που πρέπει να είναι σαφές ε, στα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να ισχύουν ίδιες προδιαγραφές όπως και στην Ευρώπη. Γιατί αν επιτρέψουμε στις εισαγωγέ να ισχύουν διαφορετικές προδιαγραφές, ε, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν προβλήματα στη δική μας ε, τη βιολογική παραγωγή. Εγώ προσωπικά φοβάμαι ότι οι καταναλωτές ε, αγοράζουν πολλές, πολλά βιολογικά προϊόντα από το εξωτερικό. Υποψιάζομαι ότι οι καταναλωτές συνδέουν τα βιολογικά προϊόντα και με συγκεκριμένες περιφέρειες. Έχουν γίνει έρευνες και δείχνουν ότι περίπου το 90% των καταναλωτών που αγοράζουν βιολογικά προϊόντα προσέχουν ε, τα προϊόντα αυτά να παράγονται σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Πρέπει λοιπόν Μάρτι να προσέξουμε έτσι ώστε να προκύψει ένας καλός κανονισμός, συνεργασία Κοινοβουλίου Συμβουλίου και παρακαλώ την Κομισιό να πλησιάσει την άποψη αυτών των δύο, γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε γρήγορα να επιτύχουμε συμφωνία. Άκουσα ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τελευταία έχουν πλησιάσει πάρα πολύ στις απόψεις τους. Δεν ζητά άλλο κανείς το λόγο. Οπότε στρέφαμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ρωτώ αν ο εκπρόσωπός θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα είμαι επιγραμματικός. Θα ήθελα απλώς να υποβάλω τρία σχόλια. Ως προς τη διαδικασία, άκουσα τον όρο επιταχύνω, ανάγκη επιτάχυσης σωστά. Πιστεύω ότι αν θέλουμε να διεκπαιρώσουμε το ζήτημα μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να επιταχύνουμε το αριθμό και άρα να αυξήσουμε τον αριθμό των συνεδριάσεων. Αυτή τη βδομάδα δεν έχουμε ούτε μία συνεδρία. Την επόμενη βδομάδα έχουμε τον τριμερή διάλογο. Καλό θα ήταν είχαν προηγηθεί και άλλοι τεχνικοί τριμερείς διάλογοι. Επιτάχυση ναι, με σεβασμό τη ποιότητα επίση, γι' αυτό χρειάζονται περισσότερε συναντήσει. Το θέμα των εισαγωγών, δεύτερο σημείο, πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την ισχύουσα κατάσταση στην Ευρώπη. Γιατί περάσαμε από το σύστημα της συμμόρφωσης που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, όλες οι ανεπτυγμένες χώρες ε, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εμείς λέμε, δεν θέλουμε να είμαστε υπερβολικά ε, ευέλικτοι και να αναζητούμε εξαιρέσεις για τις ε, εισαγωγές. Δεν είναι σωστό αυτό. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο του Φιλανδού, αν δεν κάνω λάθος, ε, Ευρωβουλευτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε αλλαγή των ισχυρών των κανόνων. Εμεί προτείναμε διατήρηση των εφισταμένων κανόνων, ούτε ζητήσαμε αλλαγή του όρου land-based σε soil-based. Σα ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγο και πάλι στον εισηγητή μα. τον κύριο Χόισλιν, παρακαλώ. Ja, liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τις ε, προτάσεις σας είναι πολύ ωραίο που θέλετε να συζητήσουμε, αλλά επισήμανα ότι έχουμε συμφωνήσει. Τώρα εγώ δεν μπορώ να λέω την προσωπική μου άποψη, ε, πρέπει να εκφράζω την άποψη του Κοινοβουλίου και θα κάνω ό,τι μπορώ, ε, παρότι σε ορισμένα θέματα είμαι διαφορετικής άποψης, φαίνεται αυτό από τις τροπολογίες. Έχω όμως μια εντολή και αυτήν θα σεβαστώ ο συνάδελφος προηγουμένως το έφηξε. η πλειοψηφία της Επιτροπής συμφώνησε ως προς το ότι πρέπει να πούμε με σαφήνεια ότι θέλουμε η γεωργία αυτή να γίνεται στο έδαφος. Υπάρχει βέβαια, σας είπα, το θέμα των θερμοκηπίων, κυρίως ας πούμε στη Βόρεια Σουηδία να συνεχίσουν αυτά ε, να λειτουργούν γιατί μπορούν να παράγουν βιολογικά προϊόντα σε γλάστρες, σε δοχεία. Τέτοιο προηγουμένω και κάποιος άλλος δεν θέλουμε μια γεωργία η οποία να ε, χρησιμοποιεί κάποιες ουσίες και μετά να χαρακτηρίζεται βιολογική αυτή είναι η ουσία του θέματος. Δεν θέλουμε αυτό να γίνεται και στα θερμοκήπια, να χρησιμοποιούν κάποια διατροφικά συστατικά που δεν είναι απόλυτα βιολογικά και μετά να χαρακτηρίζονται ε, βιολογικά προϊόντα ή βιολογικές καλλιέργειες. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε. Όσον αφορά τους ελέγχους, αποφασίσαμε να μην διατηρήσουμε τους ετήσιους ελέγχους. Αυτό βεβαίω σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε κάποιους ε, ελέγχους όταν διαπιστώνουμε κίνδυνο. Αποφασίσαμε όμως να μην έχουμε τήσιους ελέγχους και αυτό θα τηρήσω. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να αυξηθούν οι έλεγχοι εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι συντρέχει κάποιος κίνδυνος. Ο Στάλφος Ντες μίλησε για το περιφερειακό στοιχείο. Η συζήτηση θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα για την εντοπιότητα και την βιολογική παραγωγή. Αυτά τα δύο στοιχεία αυτά δεν γίνονται δεκτά από όλα τα κοινοβούλια. Μιλήσαμε για κάποια χιλιομετρική απόσταση. Το θέμα της εντοπιότητας ε, θα το εντάξουμε, αλλά αναμφίβολα. Αυτό είναι ένα θέμα που σας λέω, δεν είναι τόσο απλό. Για αυτά που είπε ο συνάδελφος Άγνιου, Εγώ δεν νομίζω ότι οι βιολογικές καλλιέργειες ε, βάζουν σε κίνδυνο την, ε, τις παραδοσιακές. Πρέπει κάπως να συνυπάρχουν όλες και στο θέμα ε, των ζυζανιοκτώνων. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι βιολογικές καλλιέργειες είναι εκείνες οι οποίες υποφέρουν από τα ζυζανιοκτώνα που και τα φυτοφάρμακα μάλλον που χρησιμοποιούν οι παραδοσιακές καλλιέργειες το θέμα των οριακών τιμών. Εκεί η στάση μας είναι καθαρή. Για μας οι βιολογικές καλλιέργειες δεν σχετίζονται με οριακές τιμές. Εμείς επιτιμούμε να ισχύει σε όλα τα επίπεδα και να βελτιωθεί η αρχή της πρόληψης. Ε, υπάρχουν κενά, θα τα δουλέψουμε, η θέση μας είναι ξεκάθαρη και νομίζω συμφωνούμε επ' αυτού με το Συμβούλιο. Μπορούμε πραγματικά εκεί να βρούμε κάποια λύση. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό, στους σπόρους υπάρχει ένας ε, κανονισμός ε, που ε, είναι ελπιδοφόρος γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι από μια ημερομηνία και μετά όλοι θα χρησιμοποιούν βιολογικούς σπόρους. Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση που είναι πιο ρεαλιστική. Πάμε τώρα στις αγωγές, γιατί έχει δύο όψεις το όλο θέμα. Ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές στις ε, εισαγωγές πράγματι δεν είναι δυνατόν να αμφισβητείτε ή να αμφισβητούνται αρχές βιολογικής καλλιέργειας, φυτοφάρμακα. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση ούτε τα ορυκτά λιπάσματα. Καμία σχέση με τις βιολογικές καλλιέργειες. Και θα αναφέρω δύο παραδείγματα όπου δεν είναι εύκολο να μεταφέρουμε τους δικούς μας τους κανονισμούς σε άλλες χώρες ακόμα και σε εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Αν πούμε ας πούμε ότι ε, οι χείροι πρέπει να παίρνουν ζωοτροφή μόνο με σανό και πάμε κάπου που δεν υπάρχει όμως αυτό το σανό δεν είμαστε δεν μπορούμε να επιβάλλουμε να γίνονται εισαγωγές σανού για να τρέφονται αποκλειστικά και μόνο με αυτές τις ζωοτροφές χείροι. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ή για το θέμα των ε, φινίκων. Εισάγουμε φινικέλαιο. Ε, δεν υπάρχουν παντού φινικές, άρα κάτι πρέπει να δούμε και δεν τι θα κάνουμε. Δεν πρόκειται ε, για τα βιολογικά προϊόντα το να καταλήξουμε στο να έχουμε απόλυτα βιολογικά προϊόντα και για να τα πετύχουμε θα σκοτώσουμε όλα τα δάση, θα τα ξεριζώσουμε. Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε ε, στο άλλο άκρο. Σας λέω λοιπόν για άλλη μια φορά με απόλυτη σαφήνεια ότι υπάρχει νομοθεσία. Δεν είναι ότι μπαίνουμε σε χαρτογράφητα νερά. Ε, απλά πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε με το να πούμε γρήγορα, γρήγορα θα συμφωνήσουμε και μετά από δύο χρονιά να επανέλθουμε στο θέμα. Πρέπει όλα αυτά να ε, είναι κάπως ε, λογικά. Υπήρξαν πάρα πολλές ε, τεχνικές συναντήσεις συναντήκαμε με τους εκπροσώπους Επιτροπής, προσπαθήσαμε να επιτύχουμε συμβασμούς και εγώ σας λέω πολύ σοβαρά ότι θα ήταν σκόπιμο κατά καιρού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδεικνύει κάποια ευελιξία και να ε, επιδιώκει συμβασμούς, όχι απλά να λέει ότι έχουμε καταθέσει την ε, καλύτερη πρόταση. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει σε αυτό το δύσκολο θέμα για αυτή την έκθεση και ελπίζω τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κυρίε και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διάταξης. Αποτελεί έκπληξη βεβαίως αυτό, αλλά έτσι ήρθαν τα πράγματα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στι 9. Παρακαλώ να θυμηθείτε να φέρετε και την κάρτα σας, γιατί θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίε. Καλό βράδυ σε όλου. και τα ξαναλέμε εδώ αύριο το πρωί στι 9. Πέρα συνεδρίασης.